οποιοδήποτε ζητήματο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ που μας ε, δίνετε την δυνατότητα να σα ενημερώσουμε για την αποστολή αυτή ε, παρατήρηση εκλογών ε, τον περασμένο μήνα. Καταρχά είχα την τιμή να ηγηθώ αυτή τη εξαμελού επιτροπή και θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στο Κυργιτστάν. Επίσης να ευχαριστήσω τη γραμματεία και το διοικητικό προσωπικό που μας βοήθησε. Το Κυργιστάν ε, θεωρείται η πιο ανοιχτή και δημοκρατική χώρα της ε, Κεντρικής Ασίας. Το Κοινοβούλιο παρατηρεί τις εκλογές στη χώρα αυτή από το 2005 και θεωρούμε ότι η χώρα αυτή είναι μοναδική περίπτωση στην περιοχή και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί. Αυτές οι εκλογές ήταν σημαδιακές διότι αφενός συνεισφέρουν στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών με ομαλή μετάβαση της εξουσίας. Οι εκλογές έγιναν υποκανονικό, ομαλό θα λέει κανείς πνεύμα πολιτικής αντιπαράθεσης ή στο τέλος ο κύριος Τζεμπέκοφ, ο πρόεδρος που υποστήριζε ο αποχωρών πρόεδρος Αταμπάγεφ, επέτυχε το μεγαλύτερο ποσοστό, ο αντίπαλος του ε, έλαβε 34,5 και η συμμετοχή ήταν 56, κάτι Ο κύριος Μπομπάνοφ ε, διαμαρτυρήθηκε για διάφορες ε, παρεκκλήσει στη διαδικασία, αλλά αναγνώρισε την ήττα του και ότι ο λαός τοποθετήθηκε και ψήφισε. Αυτό επίση ήταν θετικό και αθλητικό. Ε, μάθαμε την περασμένη εβδομάδα ότι παρετήθηκε από ηγέτη της ε, κοινοβουλευτική ομάδας αντιπολίτευσης ο κ. Μπαμπάνοφ εκκρεμούσεις και μιας ε, ποινική έρευνας εναντίον του. Τώρα, σε αντίθεση με πολλές άλλες περιοχές της Κεντρικής Ασίας, ο κύριος Αταμπάγεφ ε, σεβάστηκε τον περιορισμό της μίας θητείας, αλλά αναμένουμε να δούμε πόσο ενεργός θα είναι στο μέλλον, μια και τον αντικαθιστά ο αγαπημένος του υποψήφιος. Ο κύριος Ναζαρμπάγεφ τώρα του Καζακστάν είχε λάβει το είχε υποδεχθεί τον υποψήφιο αυτόν, το οποίο συνεισφέρει σε ένα πνεύμα, εν πάση εκτός αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Είχαμε και το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, και την ε, κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση της ε, Ολομέλειας του OSD. Έχετε λάβει σχετικά αντίγραφα των εγγράφων αυτών στα, στους φακέλους σας. Στο Μπίσκεκ ε, είχαμε συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών και Εσωτερικών, όπως και τους υπευθύνους της εκλογικής διαδικασίας, εκπροσώπους του τύπου και της κοινωνίας των πολιτών και με τους πρέσβεις μας. Ε, ε, εκεί ελάβαμε μια ενημέρωση εν ώψη των εκλογών. Την ημέρα των εκλογών στο Μπίσκεκ είχαμε τρεις ομάδες, στο Μπίσκεκ μάλλον, στο Μπελιτσί και στο Καραμπάχ, ε, καλύπτοντας διάφορες από τις περιοχές της περιφέρειας της χώρας και παρατηρήσαμε και την καταμέτρηση των ψήφων. Εμείς χαιρετίζουμε την, την πολιτική ανταγωνιστικότητα της πάντων διαδικασίες και το γεγονός ότι διεξήχθησαν ελεύθερα. Υπήρξαν κάποια σημεία που σημειώσαμε, τα οποία μας ανησύχησαν κάπως την ημέρα των εκλογών. Αυτά τα είχε θέσει ήδη ο κ. Παντσέρη πριν από την έλευσή μας στο Μπίσκεκ σχετικά με περιορισμούς που είχαν ε, επιβληθεί στον τύπο, στα μέσα ενημέρωσης το οποίο επηρέασε τον δημόσιο διάλογο που διεξήχθη και παρότι είχαν διοργανωθεί πολιτικές συζητήσεις στην τηλεόραση που συνεισφέρουν στον πλουραλισμό συνολικά δεν εδόθηκε μια ισορροπημένη και δίκαιη κάλυψη των, της διαδικασίας ε, των εκλογών. Εμείς θα θέλαμε να ενισχυθεί η διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας με αυτόν τον τρόπο. Είχαμε ακούσει και κάποιες φήμες ε, για ε, πολιτική επιρροή που ασκεί τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Το θετικό είναι ότι έχουμε μάθει για κάποιες για την εξέλιξη κάποιων ποινικών διώξεων κατά ηγετών της αντιπολίτευσης εκ μέρου του κόμματος της ε, πατρίδας, Fatherland Party, οι οποίες πολιτικές διώξεις ενδεχομένως είχαν ε, πολιτική πρόθεση και ένας από τους αρχικά υποψήφιους για την προεδρική εκλογή είχε κατηγορηθεί για συγκεκριμένα δικήματα προ των εκλογών σύμφωνα με τις αρχές της αστυνομίας εσχεδίαζε, της ασφάλειας εσχεδίαζε πραξικόπημα ο υποψήφιος αυτός. Όλες αυτές οι ανησυχίες πηγαίνουν πέρα από την στενή περίοδο της διεξαγωγής των εκλογών. Εμείς ως Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε δημοκρατική σταθερότητα στο Κυριτστάν ως τμήμα του τακτικού μας πολιτικού διαλόγου και υπό τα κίνητρα που δίνουμε για βιώσιμη και σταθερή διακυβέρνηση. Απέστειλα ήδη επιστολή στον κύριο Λάγκε, πρόεδρο της ΣΥΝΤΕ, εξηγώντα τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και τις ανησυχίες. Η σημασία των σχέσεων Κυργιστάν-Ευρακή Ένωση ε, μα εξηγήθηκε πριν από την επίσκεψη στο Μπίσκεκ, όταν στι 9 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε ότι το Συμβούλιο είχε υιοθετήσει εντολή για την ε, Επιτροπή και την είπατε εκπρόσωπο για να διαματευθεί ε, συγκεκριμένη εταιρική συμφωνία με το Κυργιστάν με κοινή δέσμευση ενίσχυσης και υποστήριξης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών και της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος όπως και της υποστήριξης της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Σύντομα θα χρειαστεί να επικυρωθεί η συμφωνία αυτή, το πλαίσιο της ανάπτυξης των σχέσεων με το Κυριστάν έχει βεβαίως ε, και το στοιχείο ότι ο βασικός στρατηγικός εταίρος είναι η Ρωσία και εκεί είναι ο βασικός εμπορικός εταίρος. Το 39% του εξωτερικού χρέους της χώρας είναι η ιδιοκτησία κινέζικης πλέον, αλλά υπάρχουν έντονα αντικινέζικα συναισθήματα στην κοινωνία από ό,τι φαίνεται. Οι σχέσεις πριν από τις εκλογές ε, μπήκαν σε μια φάση δυσχέρειας, για να το πω έτσι, Και για να ολοκληρώσω την ενημέρωσή μου, ένα μήνα πριν από την ε, εντολή διαπραγμάτευσης, τον Νοέμβριο, η κυρία Μογκερίνη επισκέφθηκε τον Μπισκέκ και επανέλαβε την συνεχή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, την, ε, για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να λάβουν χώρα στο Κυργιστάν και σχετικά με την αποστολή παρατήρησης εκλογών και εμείς λοιπόν θα πρέπει να αναλάβουμε το δικό μας ρόλο ώστε η χώρα να εφαρμόσει όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται. Ως επικεφαλής της αποστολής εγώ θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για την πλήρη αυτή παρουσίαση που μας κάνετε όσον αφορά τις εκλογές και την περίοδο μετά τις εκλογές στο Κυργιστάν. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μερνέσκο τώρα θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Δεν θέλετε το λόγο, μάλιστα δεν κατάλαβα καλά. Σας το συγγνώμη. Δεν θέλει κανείς να πάρει το λόγο από ό,τι φαίνεται, άρα μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό λέγοντας ότι η αιτήρηση αυτή η παρουσίαση μας έγινε από την κυρία Αντρικένε μας καλύπτει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική εργασία που κάνατε και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης έχουμε τη σύσταση προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΕΒ όσον αφορά την εξάλληψη των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών, στοχοθετημένη καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Θα ήθελα να εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Σχέδιο έκθεση το οποίο μας έχει ετοιμάσει ο κύριος Νάρτα, ο εισηγητής μα. Η καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία καταπολέμησης της ίδιας τρομοκρατίας και αποτελεί ένα πια από τα κομβικά σημεία του προβλήματος. Αποτελεί πολύ σημαντική πρόκληση να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καθότι οι τρομοκράτε και οι βρίσκουν πολλούς διαφορετικού τρόπους χρηματοδότηση κάθε φορά. Τα κρατη θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να μειωθεί η χρηματοδότηση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Ο κύριος ε, Νάρ, τώρα ο μας, θα μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση του σχεδίου εκθεσής του. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αναφερθώ στο σχετισμό του μακροσκοπικού με το μικροσκοπικό επίπεδο του φαινομένου της τρομοκρατίας, μιλώντας για τον τζιχαντισμό η άμεση καταστροφή της ISIS ίσως να οδηγήσει σε ένα franchise τρομοκρατίας στην οικονομική πραγματικότητα του φαινομένου. Έχοντας δει και τα κρούσματα της ε, Νίκαιας, ε, της Βαρκελόνης και του Λονδίνου. Είδαμε και σημαντικές τραπεζικές απάτες σχετικά με ε, τις προσπάθειες χρηματοδότησης των τρομοκρατικών ομάδων. Ωστόσο, πρέπει να πάμε να εξετάσουμε τις δικασίες χρηματοδότησης από τα κρυπτονομίσματα μέχρι τους ε, παραδοσιακούς τρόπους, μεθόδους πληρωμής, εμβασμάτων, μεταφορών κεφαλαίων. Έχουμε καταγράψει διάφορες παρατυπίες της διαδικασίας αυτής. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να νομοθετήσουν ώστε να ανοίξουν οι τρέχοντες λογαριασμοί χωρίς κανέναν περιορισμό για τις ε, υποεξέταση περιπτώσεις ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα περνούν με μη ρυθμισμένο τρόπο οι μεταφορές αυτές κεφαλαίων. Νομίζω ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα ρυθμίζουμε τις ε, μεταφορές αυτές, τα εμβάσματα αυτά, το οποίο δεν έχει, δεν αποσκοπεί ούτε σε, δεν έχει φορολογική πρόθεση, ούτε περιορισμού βεβαίως ε, των οικονομικών και πιστοτικών δυνατοτήτων ε, των επιχειρήσεών μας, μια και δεν μπορούμε να έχουμε και διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οικονομική μας κοινότητα, μεταξύ εμβασμάτων που μπορεί να γίνονται μεταξύ κατοίκων ή πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη κατοίκων ή πολιτών. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε την τέταρτη οδηγία κατά του ξεπλήματος του χρήματος για να διευκολυνθούν οι έρευνες ε, των ε, αρχών ε, έρευνας του οικονομικού εγκλήματος και θα επιτρέψει και στην ανταλλαγή δεδομένων γιατί έχουμε μια απολύτως ανισόρροπη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Σε πάρα πολλές χώρες μπορούμε να γνωρίζουμε ποια, ποιοι είναι οι, τρέχοντε, οι τρέχοντες λογαριασμοί που έχει οποιοδήποτε πρόσωπο, αλλά από την άλλη μεριά δεν υπάρχει ανταλλαγή των δεδομένων των σχετικών αυτών μεταξύ των κρατών μελών, το οποίο μας οδηγεί σε μια πολύ περίεργη στάση που διατηρούμε σε σχέση με τραπεζικά ζητήματα. Στις συστάσεις λέμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα και να επισημοποιήσουμε την άτυπη συνεργασία που έχουμε αυτή τη στιγμή μεταξύ ε, υπηρεσιών πληροφοριών για το χρηματοοικονομικό έγκλημα, αυτή τη στιγμή γίνεται όχι απλώς άτυπα η συνεργασία ανταλλαγή αυτή, αλλά χωρίς σταθερότητα. Και τελικώς χάνουμε ένα σημαντικό στοιχείο. Να έχουμε δηλαδή ένα κέντρο δεδομένων, το οποίο να εξετάζει την πραγματικότητα όπως είναι και όχι να εξετάζει μια ιδεατή κατάσταση. Είχαμε μιλήσει για τη δημιουργία ενδεχομένως μιας υπηρεσίας πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι απολύτως αδιανόητα στα πλαίσια της ε, κυριαρχίας που έχουν σήμερα τα κράτη-μέλη. Η προσπάθεια της δημιουργίας ενός FBI αντίστοιχου είναι απολύτως αδύνατη. Πρέπει να δουλέψουμε με αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, με τη συνεργασία ή στα όρια και τα πλαίσια που έχει αυτή τη στιγμή. Επομένως μιλούμε για τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών που υφίστανται, ώστε να έχουν ενδεχομένω ένα κέντρο δεδομένων, μια τράπεζα πληροφοριών, αν θέλετε να το πούμε έτσι, για να μπορούν να επικοινωνούν. Γιατί μπορεί ένα φιλανδικό δικαστήριο να εξετάζει μια, ένα κρούσμα τρομοκρατίας ή ένα πορτογαλικό δικαστήριο να εξετάζουν μια περίπτωση λαθρεμπορίου ναρκωτικών και να μην γνωρίζουν αυτά τα δύο δικαστήρια, αυτοί οι δύο εισαγγελεί, ότι πρόκειται για το ίδιο φαινόμενο, για την ίδια κίνηση. Αυτά τα κενά θα πρέπει να τα κλείσουμε. Δεν μπορεί να γίνεται ανενόχλητα το, να διεξάγεται το έγκλημα μπροστά στα μάτια των ε, δικαστικών λειτουργών. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που μας δημιουργεί προβλήματα. Θα πρέπει να αφήσουμε λοιπόν κατά μέρος την ανοησία θα έλεγα του πολιτικά ορθού και να προχωρήσουμε σε μια οδηγία που να αντιμετωπίζει πραγματικά τις απειλές της δημοκρατίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. ευχαριστούμε πολύ κύριε Σιγητά. Να δώσω καταρχάς το λόγο στον κύριο Γκάλερ από το ΕΛΚΑ, εξ ονόματος του κύριου Άρκουσον, που ήταν σκέδος εισηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ που ζητήθηκε από τον συνάδελφο να διαβάσω το, την, τις παρατηρήσεις του. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την έκθεση αυτή που έρθει την κατάλληλη στιγμή. Η καταπολέμηση κατά του ISIS δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο να κηρύξει πρόωρα την νίκη κατά των τρομοκρατών. Θα πρέπει ανταυτού να προσπαθήσουμε να αντλήσουμε διδάγματα και από τις νίκες και από τις ήτες της ISIS. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με την χρηματοδότηση τρομοκρατίας και πώς αυτό μπορεί να έχει οδηγήσει τελικά στην πτώση της τρομοκρατικής αυτής οργάνωσης. Δεύτερο μάθημα. Μετά τη διάλυση μιας οργάνωσης αντινάησης που είναι τόσο μεγάλη θα προκύψει ένα μεγάλο κενό. Ξέρετε ότι ορισμένοι θα κάνουν πάντο δυνατό προκειμένου να καλύψουν το κενό αυτό με νέες τζιχαντιστικές οργανώσεις και γι' αυτό θα χρειαστούν χρήματα. Και γι' αυτό το λόγο το ψήφισμα αυτό έρχεται πάλι την κατάλληλη στιγμή. Με άλλα λόγια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εντοπίσουμε και να διαλύσουμε τι χρηματοπιστωτικέ δομέ που στηρίζουν τι τρομοκρατικέ οργανώσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να διαλύσουμε τι οργανώσει αυτέ καθ' αυτές και να αποφύγουμε την μελλοντική ε, επανεμφάνισή τους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διαλύσουμε τα δίκτυα χρηματοδότησης τα οποία εφίστανται αυτή τη στιγμή για τις τρομοκρατικές αυτές οργανώσεις. Ως προς αυτό λοιπόν θα πρέπει να θυμόμαστε το ζήτημα της επιβολής και της εφαρμογής, ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, δηλαδή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών μυστικών πληροφοριών. Το Ευρωπαϊκό Λευκό θεωρεί ότι η ιδεολογία πίσω από τον τσιχαντισμό είναι ουσιαστικά μια θεοκρατική ιδεολογία που θέλει να υποτάξει όλη την κοινωνία και που προβλέπει ότι η νομοθεσία θα πρέπει να συνάδει με την Ισλαμική Σαρία. Ο σαλαφισμός λοιπόν δεν έχει να κάνει με την πνευματικότητα, αλλά σε μια πρώτη φάση έχει να κάνει με το ίδιο το δίκαιο, το οποίο θα πρέπει να ισχύει και το οποίο προφανώς εμάς μας βρίσκει αντίθετους, καθότι θεωρούμε ότι θα πρέπει θρησκεία και κράτος να είναι δύο ξεχωριστές εντελώς εξουσίες. Ξέρετε επίσης ότι πολλές φορές οι στόχοι των τζιχαντιστών ε, είναι και πολιτικής φύσης και πολλές φορές προφανώς γίνεται ένα μάγαλμα μεταξύ τζιχαντιστών και μουσουλμάνων. Το Ευρωπαϊκό Λεκοκόμμα λοιπόν θεωρεί ότι θα πρέπει να ξαναδούμε την πολιτική μας απέναντι στις χώρες εκείνες οι οποίες ε, χρηματοδοτούν τον Ισλαμιστικό, την Ισλαμιστική τρομοκρατία. Ας δούμε επίσης τι γίνεται και με την Τουρκία, καθώς επίσης και με τη διασπορά της Τουρκίας, όπου βλέπουμε ότι πολλές φορές η δράση της γίνεται πάρα πολύ ανισχυτική. Ενδεχομένω και αυτό θα πρέπει να αναφερθεί. Το ΕΛΚ θεωρεί ότι οι αρχέ των κρατών μελών θα πρέπει να παρακολουθούν τη χρηματοδότηση από ξένε οντότητε για τζαμιά και Ισλαμικού συλλόγου και ότι θα πρέπει να προβλέπεται απαγόρευση τέτοιες χρηματοδότησης κάθε φορά που έχουμε εύλογους λόγους να πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη χρηματοδότηση της βίας ή ακόμα και της τρομοκρατίας στις χώρες μας. Βάσει όλων αυτών, Είμαι σαφώ υπέρ τη έκκληση που γίνεται προ τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσουν ένα σύστημα παρακολούθηση προκειμένου τα τσαμιά οι πολιτισμικοί οργανισμοί και άλλες οντότητες θα πρέπει να κοινοποιούν όλα τα στοιχεία για τη χρηματοδότησή τους και για τα κεφάλαια που φτάνουν αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να δούμε τι θα γίνεται με το σύστημα αυτό της Χαβάλα, Χαβάλα που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως άτυπη μεταφορά κεφαλαίων για να χρηματοδοτηθούν τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να είναι σαφή η διατύπωση στο κείμενο για το σύστημα αυτό. Ο εισηγητής επίσης θα μπορούσε να αφαιρθεί λίγο στο μέγεθος που έχει το πρόβλημα αυτό στην Ευρώπη, γιατί το σύστημα Χαβάλα δυστυχώς δεν έχει ακόμα απασχολήσει ιδιαίτερα την όλη συζήτηση που έχει γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τέλος του κειμένου γίνονται διάφορες προτάσεις για νέες νομοθεσίες. Πώς πιστεύετε ότι μπορούν αυτές να διευθυντηθούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Προσβλέπουμε πάντως και στη μελλοντική συνεργασία που θα έχουμε με τον εισηγητή και τον ευχαριστούμε μέχρι στιγμής για τη σημαντική εργασία που έχει κάνει. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος ε, περισσότερο στα από προφορικά. Μετά περνάμε στους σοσιαλδημοκράτες και έχουμε και τον κύριο Λίτς εξ ονόματος ε, του σχεδόν Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ δεχτείτε την συγγνώμη για την απουσία μου. Πρόκειται για ένα καλό σχέδιο έκθεσης. Οι συζητήσεις που έχουμε ξεκινήσει έχουν στόχο να δουν μέτρα που θα λειτουργήσουν στην πράξη κάθε σύσταση θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά. Υπάρχουν θετικές διατυπώσεις ε, για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας και πρέπει να τονίσουμε ότι σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα πρέπει να φροντίσουμε ότι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε δεν θα αποξενώσει ομάδες ή θα χρησιμοποιήσει στερεότυπα γύρω από το Ισλάμ. Ήδη είχαμε επικοδομητικές ε, συζητήσεις ε, όπως ε, παραδείγματος χάρη την πρόταση για κυρώσεις σε όσους εμπορεύονται με το ΝΤΑΕΣ αλλά και βεβαίω το πώς μπορούμε να σταματήσουμε το εμπόριο αρχαιοτήτων και πολύτιμων λίθων που χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και αναμένω την περαιτέρω συζήτηση επί του θέματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ομάδα σας που ήσασταν και σύντομοι. Περνάμε λοιπόν στον κύριο Φανόρντεν από το ΕΣΥΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ τον Χαβιέ. Μια εξαιρετική βάση για μια έκθεση. Νομίζω μας αρέσει η γενική κατεύθυνση και το γεγονός βεβαίως ότι κοιτάει προς τα έξω. Πρώτα απ' όλα κάτι το γραφειοκρατικό. Έχω μια ερώτηση για την δομή της έκθεσης που είναι κάπως πρωτότυπη. Έχω πρόβλημα με τις πρωτοτυπίες, αλλά δεν ξέρω αν βοηθάει στην συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί η παράγραφος 1 είναι όλη η έκθεση ουσιαστικά. Νο, κανονικά, στις εκθέσεις μας έχουμε διάφορες παράγραφους. Ο πρόεδρος. Ε, είναι σύσταση γι' αυτό. Δεν είναι μια παραδοσιακή έκθεση. Μάλιστα, ωραιότητα. Ωραία λοιπόν. Ακόμα και έτσι. Επίσης υπάρχει μια διάκριση που πρέπει να γίνει μεταξύ αυτού του οποίου θα έλεγα χρηματοδότηση των διεθνών τρομοκρατικών οργανώσεων όπως το Ισλαμικό κράτος, η Αλκάιντα κτλ. και η χρηματοδότηση που έρχεται στις χώρες μας για να προωθήσει την τρομοκρατία. Μπορούμε να το πούμε, θα έλεγα, την προτζιχαντιστική φάση, την ριζοσπαστικοποίηση δηλαδή και οι πηγές της χρηματοδότησης για τους για τα Αμερικίνα, τζαμιά ή μετρεσέδε που προωθούν την ακραία ιδεολογία. Είναι βεβαίω ε, διαφορετικά ένα, αλλά σχετιζόμενα ζητήματα. Και πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση. Μιλήσατε για την ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχει βεβαίως τέτοια ανταλλαγή πληροφοριών και να έχετε κατά νου ότι υπάρχει και μια ομάδα δράσης ε, θα το ξέρετε που συστάθηκε το 1989 μετά από πρωτοβουλία των G7, αλλά τώρα έχει μέλη διάφορες χώρες ανά τον κόσμο που προσπαθεί να θέσει κάποιες προδιαγραφές για πράγματα όπως το ξέπλυμα χρήματος, καταπολέμηση της, ε, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ε, φαίνεται ότι έχει, ε, έχει κάποια σχέση με το αντικείμενο σας, αλλά δεν βλέπω κάποια αναφορά είμαι κάπως επιφυλακτικός για οτιδήποτε λέει ότι πρέπει να υπάρξει ακόμα κάτι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει στήριξη για μια υπηρεσία πληροφοριών της Ένωσης και δεν ξέρω αν αυτό εννοείται. Νομίζω ότι εννοείται μια πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών. Έχουμε μια πλατφόρμα ήδη στην Europol. Και κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι βεβαίως έχουμε την Ειδική Επιτροπή για την Τρομοκρατία που εξετάζει πολλές πτυχές ε, του προβλήματος αυτού και μια πτυχή που εξετάζουμε συγκεκριμένα είναι η χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατίας. Πρέπει λοιπόν ε, να δούμε ότι υπάρχει αυτή η επιτροπή. Αυτά θα θα τα βάλουμε και σε τροπολογίες, αλλά είναι μια εξαιρετική έκθεση με αρκετά καλά πράγματα και θα προσπαθήσουμε να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ μου. Ο κύριος Μπούκνερ τώρα για τους πράσινους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή την πολύ καλή έκθεση, μια πολύ σημαντική αφετηρία. Συμφωνώ και με αυτό το οποίο, με αυτό το οποίο είπε ο προλαλής Το σημαντικότερο θέμα είναι ότι δεν αρκεί να δούμε τις χρηματικές ροές που πάνε απευθεία στις τρομοκρατικές οργανώσεις, γιατί στο παρελθόν, παραδείγματος χάρη, είχαμε την πώληση πετρελαίου ή έργων τέχνης που ήταν ε, λάφυρα, κλεμμένα. Οπότε πρέπει να επεκτείνουμε το πεδίο εδώ Και υπάρχουν κάποιες ε, χρηματοοικονομικές μέθοδοι που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Κάτι τα λοιπά. Συμφωνώ πλήρως με τους προλαλήσαντες. Ευχαριστώ. από το EFDD, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σίγουρα η έκθεση αυτή είναι πολύ καλή και θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε πολλά σημεία σε σχέση με αυτά που ο κύριος Γκάλερ πριν από λίγο, μιλώντας εξ ονόματος του κυρίου Αντάκτουσον, χρηματοδότηση για τα τζαμιά και παρακολούθηση της χρηματοδότησης αυτής και των κεφαλαίων αυτών που διοχετεύονται προς τα τζαμιά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι εθνικέ υπηρεσίε πληροφοριών λειτουργούν ήδη πολύ καλά. Ο Τζέφρι Βανόρντεν μα είπε ότι ήδη υπάρχει και η Ιντερπολ και η Ευρωπόλ, αλλά και μια ομάδα δράση η οποία συντονίζει τι εθνικέ αρχέ μυστικών πληροφοριών. Ξέρετε επίση ότι στα πλαίσια της ΕΙΕΔ έχει γίνει και μία ανοιχτή συζήτηση και αυτό έγινε και πριν το δημοψήφισμα για το Brexit για το πώς θα μπορούσαν να ενδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο οι εθνικές υπηρεσίες και μεταξύ τους συνεργασία, οι εθνικές υπηρεσίες μυστικών πληροφοριών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι η συνεργασία αυτή και με το Μένο Βασίλειο θα συνεχιστεί και μετά το Brexit. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τώρα ότι όντω η ISIS προσπαθεί να ανασυσταθεί, να αναδιοργανωθεί και σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Αφρική. Είπατε επίση ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε τις πιστοτικές κάρτες και τις σχετικές συναλλαγές. Ας μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί όμως τρομοκράτες βρίσκονται εκτός τραπεζικού συστήματος και θα συνεχίσουν να βρίσκονται εκτός τραπεζικού συστήματος. Όσον αφορά τις ανησυχίες για την Χαουάλα, θεωρούμε ότι όντω θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, αλλά αν κάνουμε τα όσα προτείνονται στην έκθεση αυτή, δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Πάρα πολλοί χρησιμοποιούν την άτυπη αυτή μεταφορά κεφαλαίων απλώς για να κάνουν ε, ε, εμβάσματα, κυρίως ε, μεταξύ μελών μιας οικογένειας. Νομίζω ότι δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα, να ακολουθήσουμε τα όσα λέγονται στην έκθεση αυτή για την αντιμετώπιση της Χαουάλα. Τώρα, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών. Νομίζω ότι αυτό όμω ε, ήδη έχει γίνει. Οι ε, υπηρεσίες μυστικών υπηρεσιών εν γέννη συνεργάζονται μεταξύ τους, πετυχαίνουν θετικά αποτελέσματα. Εμείς ακούμε κυρίως τις αρνητικές ειδήσει, αν θέλετε. Έχουν καταφέρει όμως να πετύχουν πολύ σημαντικά επιτεύγματα όσον αφορά την μείωση και την εξάλληψη των πηγών εσόδων για, το, ε, για τη δημοκρατία. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αφάζερ, εξ του ΙΕΝΕΦ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμεί ε, χαιρετίζουμε την πολύ καλή αυτή έκθεση. Θα ήθελα να θέσω όμω κάποια ζητήματα ουσία. Πώ είναι ποτέ δυνατόν μόνο το 2% του βρώμικου αυτού χρήματος τελικά να εντοπίζεται. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα το οποίο θα πρέπει να θέσουμε. Πώς είναι επίσης δυνατόν στο όνομα της τρομοκρατίας και της νομοποίησης εσόδων οι τράπεζες να καταφέρουν τελικά οι τράπεζε ε, ελέγχουν τελικά όλο και περισσότερο την κοινωνία και του ίδιου του πολιτικού, Ο ίδιο ε, υπέφερα σε τέτοιο βαθμό που ενημέρωσα πρόσφατα τον κύριο Ταγιάννη λέγοντα του δεν ήμουν σε θέση πλέον να εκτελέσω σωστά την εντολή μου. Θα σας πω για ποιο λόγο έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτή την κατάσταση. Πέρα και πίσω από τη χρηματοδότηση και την νομοποίηση παράνομων εσόδων, οι πρώτοι που εμπλέκονται τελικά είναι τα κράτη και οι μυστικές υπηρεσίες τους. Ενδεχομένως θα έπρεπε εκεί να γίνει μια έρευνα, να δούμε τι κάνουν ορισμένες τράπεζες οι οποίες δημιουργήθηκαν α, για την νομοποίηση παράνομων εσόδων, όπως και ο αρμόδιος επίτροπος άλλωστε είπε. Στην Ινδοκίνα χρησιμοποιούσαμε εμείς χρήματα μια συγκεκριμένη τράπεζα προκειμένου να καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε μυστικέ υπηρεσίε και αποστολέ. Αυτό έγινε και στο Αφγανιστάν και ουδέποτε είχαμε τέτοια διακίνηση ναρκωτικών ε, όσο από τότε που αρχίσαμε πραγματικά να έχουμε εμεί δυτική παρουσία στο Αφγανιστάν. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα και να συντοπίσουμε τελικά ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες τράπεζες οι οποίες μέσω της δράσης τους προσπαθούν να ελέγξουν και τις κοινωνίες μας και τους πολιτικούς μας. και που προσπαθούν τελικά να ελέγξουν το σύνολο του οικονομικού συστήματος χωρίς να υπάρχει βέβαια κανένα αποτέλεσμα όσον αφορά την πάταξη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Θέτω λοιπόν το ακόλουθο ερώτημα. Για παράδειγμα γνωρίζουμε πάρα πολύ ότι στη Μάλτα ε, όπου έγινε και μια δολοφονία, υπήρχε μια, ένα ολόκληρο παρακλάδι τη αλβανική μαφία που ξέπλυνε εκεί πέρα χρήματα. Τι έγινε στη Μολδαβία, τι έγινε στο Μαυροβούνιο. Στη Μολδαβία χάθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ, εξαφανίστηκαν εκεί πέρα, μπορώ να πω. Αντί να ασχοληθούμε με τα ζητήματα αυτά, ασχολούμεθα με άλλε δεπτομέρειε. Ασχοληθούμε με την ουσία λοιπόν του προβλήματο. Δεύτερη ομάδα ερωτημάτων και παρατηρήσεων. Θα είμαστε πραγματικά πιο αποτελεσματικοί αν συνεργαστούμε πανευρωπαϊκά. Μα νομίζω ότι ήδη υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Χρειαζόμαστε πάλι μια νέα υπηρεσία, ένα νέο οργανισμό για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Δεν νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντανζό από το ΕΛΚ έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι η έκθεση είναι πολύ καλή. Συγχαρητήρια λοιπόν στον κύριο Νάρτα. Δύο σημεία θέλω να θίξω. Γίνεται μεγάλη αναφορά στο Ισλαμικό κράτος και στον Ταέσα στην έκθεσή σας. Κάθε φορά που μιλάμε όμως για τζιχατιστική τρομοκρατία θα πρέπει να ξεχνάμε και την Αλκάιντα η οποία παραμένει η πιο καλά δομημένη οργάνωση αυτή τη στιγμή, μολονότι μπορεί να μην είναι τόσο εντυπωσιακή δράση της ε, επί του παρόντος. Θεωρώ ότι το σύστημα χρηματοδότησής της είναι πολύ πιο πολύπλοκο και προηγμένο από ότι το σύστημα χρηματοδότησης για το Ισλαμικό κράτος. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει ε, να μην αφήνουμε εκτός έκθεσης ε, την Αλκάιντα, η οποία όπως σας είπα είναι, εξακολουθεί και είναι πάρα πολύ ισχυρή και πολύ ισχυρή οικονομικά και όσον αφορά το σύστημα χρηματοδότησής της. Και ξέρετε ότι κατάφερε μέσω όλων αυτών των ομήρων και των λίτρων που χρησιμοποιούσε να συγκεντρώσει τεράστια ποσά, τα οποία χρησιμοποίησε προφανώ στη συνέχεια για να χρηματοδοτήσει τη δράση τη. Πρώτον αυτό λοιπόν, όσον αφορά την Αλκάιντα. Δεύτερον, Όσον αφορά τη διατύπωση που χρησιμοποιείται, όσον αφορά τις εξηγήσεις επίσης, ο κύριος Νάρτα πολύ επιδέξια αποφεύγει την παγίδα στην οποία αναφέρθηκαν κάποιοι συνάδελφοι του να δημιουργηθεί ένας οργανισμός, επιπλέον οργανισμός. Ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι υπέρ της προστιθέμενης αξίας της επιπλέον Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας. Ο κύριος Νάρκ λοιπόν δεν μιλάει για νέα υπηρεσία οργανισμού, αλλά μιλάει για πλατφόρμα προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες είναι οι πλέον αρμόδιες για να κάνουν την εργασία αυτή. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία έγκυται στην εναρμόνιση των δικασιών και στην καλύτερη δόμηση των, της ανταλλαγής πληροφοριών, έτσι ώστε κάθε κράτος μέλος να μπορεί να συμβάλλει στην πλατφόρμα αυτή που θα δημιουργηθεί. Θεωρώ για παράδειγμα ότι η Ιταλία με την Guardia τη Finanza που έχει ήδη εργάζεται πάρα πολύ καλά για τα ζητήματα αυτά, την υπηρεσία καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος. Νομίζω λοιπόν ότι δεν έχουμε ανάλογες δυνατές αρχές ε, σε κάθε κράτος μέλος. Νομίζω ότι πρώτα θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο να έχουμε την απαραίτητη νομοθεσία, την απαραίτητη δομή και αρχιτεκτονική, προκειμένου να έχουμε εθνικές υπηρεσίες καταπολέμησης της χρηματοδότησης, της τρομοκρατίας, πρωτού ασχοληθούμε με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κυρία Γκόμες τώρα από τους σοσιαλιστές έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Στο συγγνώμη, Πρόεδρε. Πρέπει να φύγω σε δύο λεπτά, γιατί πρέπει να πάω στην Σόφια και με περιμένει το αεροσκάφος. Στο συγγνώμη. Να πω απλώς εγώ στον Χαβιέ Νάρτ ότι δουλεύουμε στην πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση των, της νομιμοποίησης των εσόδων. Η δουλειά μπλοκαρίστηκε την περασμένη εβδομάδα από το Συμβούλιο, διότι το Συμβούλιο δεν σοβαρολογεί για την καταπολέμηση του ξεπλήματος και της χρηματοδότησης της θερμοκρατίας. Όλα αυτά ενεργοποιήθηκαν από την επίθεση των Πατακλάν και τις προπληρωμένες κάρτες, αλλά τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά. Το, τα κρυπτονομίσματα είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και πρέπει να μιλήσουμε και για την Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και πολλά άλλα. είναι σημαντικό να εστιασιζόμαστε και στην τοποθέτηση του Επιτρόπου Μοσκοβισή την πρόσφατη ότι οι απάτες ΦΠΑ λαμβάνουν χώρα και απορρέουν σε περί τα 5 δις χρηματοδότησης προς τα τρομοκρατικές οργανώσεις συμπεριλαμβανομένης της Αλκάιντα Απάτες που δεν αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Χωρίς να μιλήσουμε για τις απάτες ειδικού φόρου κατανάλωσης, Σε οποίες αναφέρει και η Europol και οι οποίες έλαβαν χώρα στη Βουλγαρία από πλευρά της ISIS ώστε να κινητοποιήσει, ώστε να λάβει τελικώς περί τα δέκα δις Ας μην μιλούμε λοιπόν για προπληρωμένε κάρτες και να ξεχνούμε αυτά τα μεγέθη. Επίσης, το ρευστό, το ρευστό που μεταφέρεται σε ιδιωτικά αεροσκάφη που δεν καλύπτονται οι ρίστε των από την BNR και σε διάφορα αεροδρόμια των κρατών μελών, ιδιωτικά και μη και να συμφωνήσω ότι εξετάζοντας την προχρηματοδότηση της ε, τρομοκρατίας αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και μιλούμε για τη χρηματοδότηση τζαμιών, σχολών, σχολείων, διαφόρων άλλων φορέων. Thank you. Uh, we will continue to debate... Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος τη απουσία του εισηγητή, γιατί γνωρίζουμε ότι έχει αξιολογότατο προσωπικό και βοηθούς. Είναι πολύ κρίμα βέβαια για το επόμενο ομιλητή στον κατάλογο είμαι εγώ. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα διαβιβαστούν τα σχολιά μου στον εισηγητή. Και δίνω στον εαυτό μου το λόγο, λέει ο πρόεδρος. Δεν θα μακρηγορήσω. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον εισηγητή για την ε, γνωμοδότησή του απολύτως επίκαιρη με τα κρούσματα τρομοκρατίας που έχουμε, ώστε να παρακολουθούμε τη δίωδο χρηματοδότηση των τρομοκρατικών ομάδων. Ευχαριστώ τον ε, κύριο Νάρτ. Υπάρχουν μια-δύο περιοχές επί των οποίων σημεία, επί των οποίων θα πρότεινα τροπολογία. Καταρχά, ε, μιλούμε όλο και περισσότερο για επιθέσεις μοναχικών λύκων ή ενεργοποίηση κυτάρων, ριζοσπαστικοποίηση, με συγχωρείτε, και τα βλέπουμε αυτά σε πυκνοκατοικημένε περιοχές, νυχτερινέ επιθέσεις και άλλες επιθέσεις με αρκετά πρωτόγωνο υλικό και φθηνό στο χειρισμό του και στην αγορά του. Επομένως θα πρέπει να καλύψουμε και αυτή την τάση νομίζω στην έκθεση. Καταλαβαίνοντας ότι η εστίαση των, των τρομοκρατών δεν είναι απλώς της χρηματοδότησης, δεν είναι αυτά που τους επιτρέπουν να δρουν, έχουν μια, αν θέλετε, ιδεολογία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η εκθέση αυτή και συμφωνώ με τα σχόλια του συναδέλφου ότι πρέπει να είμαστε συνολικοί εδώ στην εξέτασή μας, πλήρης, να συμπεριλάβουμε και τη χρηματοδότηση όχι μόνο των επιθέσεων αλλά και άλλων φορέων συμπεριλαμβανομένων τζαμιών και σχολείων κτλ. Όλα αυτά που επιτρέπουν, αν θέλετε, τη ριζοσπαστικοποίηση σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πεδίο. Πρέπει να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Και το τελευταίο που ήθελα να αναφέρω είναι ότι πρέπει να έχουμε μια ολιστική, όπως λέμε, προσέγγιση και πρέπει να χρηματοδοτούμε έργα και προγράμματα που έχουν επιτυχία στις επιδόσεις τους για την καταπολέμηση της δημοκρατίας. Πρωτοβουλίες που θα είναι σε θέση να πλήξουν το θεματολόγιο της τρομοκρατίας. Είμαι ένας από τους ε, καλύτερους μαθητές γιατί τήρησα το χρόνο και θα δώσω το λόγο τώρα στον τελευταίο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα η έκθεση αυτή αποτελεί καταπληκτική βάση προκειμένου να καταφέρουμε να ενισχύσουμε λίγο περισσότερο τα μέσα τα οποία έχουμε για να καταπολεμήσουμε τη χρηματοδότηση τη ε, τρομοκρατίας. Μέσα τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μια στιγμή που εντείνεται η δράση των ε, αλλοδαπών μαχητών. Πρέπει λοιπόν να μειώσουμε τις πηγές τους, τις πηγές χρηματοδότησής τους, οι οποίοι, ε, πηγές χρηματοδότησης των τρομοκρατών που βάλουν κατά των κοινωνιών μας και των πόλεων μας. Παρ' όλα αυτά παραμένουν κάποια σημεία από των οποίων πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και να επιμείνουμε λίγο περισσότερο. Το ζήτημα της Χαουάλα, ένα ζήτημα το οποίο μας είχε απασχολήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά τζαμιά και ισλαμικά κέντρα σε πολλές χώρες, αρχή γενομένη από τη δικιά μου, όπου ουσιαστικά δεν γίνεται ο απαραίτητο έλεγχο, Δεν ξέρουμε τελικά ούτε τι διδάσκουν εκεί πέρα, ούτε τι λένε, ούτε ακριβώ κάνουν. Ξέρετε ότι η διδασκαλία γίνεται στα αραβικά, οι περισσότεροι αστυνομικοί δεν είναι σε θέση καν να καταλάβουν, να εντοπίσουν ε, ρητορική μίσους ή άλλα τέτοια στοιχεία. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε λίγο περισσότερο τη χρηματοδότηση των Ισλαμικών αυτών κέντρων και των τζαμιών που έχουμε στις χώρες μας. Ξέρετε ότι πολλά από τα κέντρα αυτά συγκεντρώνουν πάρα πολλά χρήματα τα οποία μπορούν να διοχετευτούν στη συνέχεια σε τρομοκρατικές ενέργειες. Ξέρετε ότι όταν ε, τα τζαμιά βρίσκονται υπό τον έλεγχο οργανώσεων που ε, ε, καταλήγουν να έχουν τελικά τρομοκρατική δράση, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι απουσιάζουν τελικά οι έλεγχοι αυτοί όσον αφορά την χρηματοδότηση όχι μόνο των Ισλαμικών, Ισλαμιστικών οργανώσεων, μαφιόζικων οργανώσεων, αλλά και των οργανώσεων εκείνων που πραγματικά ελέγχουν την παράνομη διακίνηση των μεταναστών. Α μην ξεχνάμε ότι μέσω τη παράνομη αυτή διακίνηση των μεταναστών έχουμε μία ακόμα πολύ σημαντική πηγή χρηματοδότηση τη τρομοκρατία και των τζιχαντιστών. Τα δύο αυτά ζητήματα λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε από κοινού και σίγουρα θα πρέπει να βαθύνουμε πολύ περισσότερο. Ως προς τα υπόλοιπα σημεία νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα θίξουμε και στην ε, συνέχεια, τα bitcoin για παράδειγμα και επίσης ε, τα έσοδα εκείνα τα οποία προκύπτουν από το εμπόριο αρχαιολογικών ευρημάτων ε, που όπως ξέρετε πάρα πολύ συχνά αποτελούν αντικείμενο παράνομης διακίνησης και πώλησης μέσω παράλληλων ε, δικτύων λαθρεμπόρων. Αλλά αυτό τέλος πάντων μπορεί να μας απασχολήσει λίγο αργότερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε με τους ομιλητές για αυτό το θέμα. Να σας πω το τι θα γίνει τώρα. Προθεσμία για τροπολογίες 21 Νοεμβρίου. 27 Νοεμβρίου, με συγχωρείτε, 11 η ώρα. 23 Ιανουαρίου θα τις επανεξετάσουμε και θα ψηφίσουμε την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου. Έτσι έχει το πρόγραμμα. Ε, ευχαριστώ τον εισηγητή και τους συναδέλφους. Ένα θέμα έχει απομείνει η ανταλλαγή απόψεων με την Αφρική και προκλήσεις για τον 21ο αιώνα. Α, ήρθανε. Μάλιστα. Πέντε λεπτά να καθίσουν και συνεχίζουμε λοιπόν με το τελευταίο θέμα. Καθίστε συνάδελφοι, ένα μικρό διάλειμμα πέντε λεπτών και συνεχίζουμε.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 Συνάδελφοι, να με το τελευταίο σημείο τη σημερινή διάταξη. ανταλλαγή απόψεων, Αφρική, προκλήσεις και ευκαιρίες για τον 21ο αιώνα. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τους καλεσμένους μας για το επόμενο θέμα που αφορά την Αφρική. Όπως ξέρετε, αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα Αφρικής ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια πρωτοβουλία του Πρόεδρου Ταγιάννη πριν από την πέμπτη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωση Αφρικής. Υπάρχουν διάφορα γεγονότα και εκδηλώσεις ε, που αφορούν την Αφρική. Υπάρχει μια διάσκεψη υψηλού επίπεδου που θα λάβει χώρα στις 22 του μηνός το απόγευμα ε, με από τις ε, ε τράπεζες μας αφορά όλους καθώς αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια και την δημοκρατία και την ε, χρήστη διοίκηση έχουμε σήμερα τρεις διακεκριμένους ομιλητές. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Όμο Αγκέκε από την Ιγυρία, βουλευτή. Καλώς ήρθατε και τον κύριο Άμπροζη, ο οποίο είναι περιφερειακός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και αναμένουμε τον κύριο Κνόντο Ντάν, τον πρόεδρο του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου. Επίσης, να καλωσορίσω τις αντιπροσωπείες από το, τα κοινοβούλια Τινησίας Μαρόκου και Νιγηρίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. σημερινή συνεδρία θα μας δώσει την ευκαιρία να συζητήσουμε ευρύτερα ζητήματα για την Αφρική. Η Ήπειρος έχει τεράστιες δυνατότητες οικονομικής και ανθρώπινης ανάπτυξης. Επίσης γνωρίζουμε ότι η Αφρική αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Ε, θέματα χρηστής διοίκησης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βεβαίως συζητήματα μετανάστευση όχι μόνο προς την Ευρώπη αλλά και ενδοαφρικανική μετανάστευση. Το φαινόμενο αυτό είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα της ανάγκης ε, η διεθνής κοινότητα, οι χώρες της Αφρικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση να οργανώσουν την συνεργασία τους για να βρεθεί μια παγκόσμια λύση για τα επόμενα χρόνια. Θέλουμε να ακούσουμε λοιπόν την αφρικανική σκοπιά για το μέλλον της Υπήρου, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεισφέρει στην διαδικασία. Θα θέλαμε να δούμε περισσότερο τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής και τον ρόλο της διεθνούς κοινότητας για την περαιτέρω ανάπτυξη της Αφρικής χωρίς άλλη καθυστέρηση. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον γερουσιαστή Όμο Αγγέγγε. Ε, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Δέκα λεπτά έχει ο καθένας στην διάθεσή του. Έχετε τον λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ. κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, εξοχότατοι συνάδελφοι Αφρικανοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι, είμαι ο Όβιε Όμο Αγγέγκε, γερουσιαστής της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της ε, Νιγηρίας, αντιπρόεδρος ε, της Επιτροπής Χερσαίων Μεταφορών, αντικαθιστώ σήμερα τον πρόεδρο Ισάνη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής εξωτερικού χρέους. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως για την ε, Αφρική ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την τιμή που έχω να σας απευθύνω τον λόγο σήμερα και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου αν πω ότι το φόρμα αυτό είναι μια πολύ, ένα πολύ καλό βήμα για να ενισχύσουμε τις σχέσεις των δύο επίρων μας. Να θυμόμαστε ότι σε κάθε δημοκρατικό σύστημα θα πρέπει ε, να γνωρίζουμε βεβαίω ότι το θεσμικό εκείνο όργανο το οποίο είναι πιο κοντά στους πολίτες είναι το Κοινοβούλιο και άρα η επαφή των κοινοβουλίων των υπήρων μας έχει μεγάλη σημασία για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής μας. Και τη στιγμή κατά την οποία οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης, ε, φυγόκητρες ε, και κεντρομόλες ε, ασκούν μια πρωτοφανή πίεση στις χώρες του κόσμου τα κοινοβούλια ως γνησιότερη έκφραση της θέλησης των λαών πρέπει να ανταποκριθούν στα προβλήματα της εποχής μας, προτείνοντας ιδέες για το μέλλον. Έτσι ακριβώς θα ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας για το θέμα αυτό, για τις προκλήσεις και ευκαιρίες του 21ου αιώνα. Είναι ε, κοινώς γνωστό πως αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της Αφρικής. Επέλεξα να εστιάσω σε αυτό, καθώς ε, κατά την άποψή μου πρόκειται για το θέμα γύρω από το οποίο περιστρέφονται διάφορα άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η τεχνολογία, το χρέος, οι υποδομές, ε, για να αναφέρω μόνο λίγα. Και βεβαίως ε, η Αφρική τις τελευταίες δεκαετίες έχει ακολουθήσει διάφορα, πολλά και διάφορα πρότυπα ανάπτυξη ακόμα βεβαίως και η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς έχουν κάνει, έχει κάνει λίγα πράγματα για να βελτιώσει την κατάστασή μας. Μάλιστα οι περισσότερες αναπτυξιακές πολιτικές δεν αντιμετωπίζουν τα θεμελιώδη ζητήματα της Αφρικής και οι αναπτυξιακές πολιτικές είναι αντιδημοφιλείς και δεν γίνονται δεκτές ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες όπου χρησιμοποιούμε τα γνωστά κλισέ όπως ε, οικονομική διαφοροποίηση, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μετασχηματισμός της γεωργίας, ε, χρηστή διοίκηση και βεβαίως το γενικότερο πλαίσιο της ε, πολιτικής το οποίο θα πρέπει να έχει ως στόχο κάποια στοχευμένα αποτελέσματα. Όλα αυτά βεβαίως όταν έρχονται σε επαφή με την πραγματικότητα της αφρικανικής πολιτικής ε, είναι σαφές το γιατί δεν έχουν αποτελέσματα. Όπως όλοι γνωρίζουμε η βιώσιμη ανάπτυξη είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχει σταθερότητα στον προγραμματισμό αντί για μια προσέγγιση ad hoc. Γι' αυτό οι ανάγκες της Αφρικής ακριβώς καθορίζονται από τις προκλήσεις αυτές στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και βεβαίως ε, το βασικό ζήτημα είναι το τι θα είναι ο κινητήρας της ανάπτυξης και πώς θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτό δεν απαιτεί να επανεφεύρουμε τον τροχό. Αντιθέτως, στη σχετική βιβλιογραφία βλέπουμε ότι έχουν γίνει ήδη πάρα πολλά από πανεπιστημιακούς, ε, πολιτικούς, ε, μεγιστάνες, επιχειρηματίες. Παραδείγματος χάρη το εμπόριο τώρα θεωρείται κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης ε, και όσοι ασκούν κριτική βεβαίως αποδέχονται ότι το εμπόριο είναι βασικό συστατικό της ανάπτυξης ταυτόχρονα με τον ίδιο τρόπο. Και τα θεσμικά όργανα περιφερειακής ολοκλήρωσης ε, θεωρούνται το κλειδί βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Αφρικής ε, και βεβαίως επέκτασης των ορίων των αγορών της. Με την αδειά σας τώρα θα ήθελα να περάσω στις προκλήσεις και ευκαιρίες για το εμπόριο στην Αφρική και θα έλεγα ότι αυτό το οποίο απαιτείται στο μέλλον είναι ένας ανασυνδυασμός ε, των ζητημάτων αυτών εμπορίου και περιφερειακής ολοκλήρωσης, τα οποία συχνά τα βλέπουμε κάπως επιφανειακά. Το εμπόριο αποτελεί καταλήτη της οικονομικής ανάπτυξης ανά τον κόσμο. Η Αφρική και η Ευρώπη έχουν ισχυρούς δεσμούς ε, και περνάμε από τις διμερείς της πολυμερείς εμπορικές σχέσεις. Όλοι βεβαίως ε, θυμόμαστε ότι έχουμε το σύστημα προτιμησιακών εμπορικών σχέσεων που περιλαμβάνει 70 χώρες της συμβάσεις ΛΟΜΕ που ό,τι και αν λένε όσοι ασκούν κριτική ήταν πάρα πολύ σημαντικές για την κοινωνική ανάπτυξη των χώρων αυτών και βεβαίως ε, και για την πρόσβαση στις αγορές. Από το 2000 όμως ε, και μετά οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των Αφρικανικών χωρών και της Νιγηρίας. Και έτσι έχουμε μια αύξηση των δυσχεριών που αντιμετωπίζει η Αφρική στο διεθνές εμπόριο, καθώς το μερίδιό της ε, στο παγκόσμιο εμπόριο μένει σταθερό και μειώνεται. Και, ακόμη χειρότερο, οι προοπτικές μετασχηματισμού των αφρικανικών οικονομιών υπονομεύονται. Θα ήθελα τώρα, κυρίε και κύριοι, να αναφερθώ στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αφρική για να υπάρξει κάποια ανάπτυξη και κατασκευή προϊόντων σε περιφερειακό επίπεδο όπως όλοι γνωρίζουμε. Οι αφρικανικές οικονομίες είναι σε γενικές γραμμές εξωστρεφής. Επιπλέον έχουμε ακριβώς την έλλειψη συμπληρωματικότητας των διαφόρων κλάδων της οικονομίας. Σχεδόν όλες οι χώρες είναι παραγωγή πρωτογενών προϊόντων και πρέπει να υπάρξει επενδύση και στις ε, τεχνολογίες και διαφορετικά είμαστε ευάλωτοι στην εκμετάλλευση από δυνάμεις εκτός της Αφρικανικής Υπήρου. Όλα αυτά βεβαίω οδηγούν σε μια αποφασιστικότητα για την ολοκλήρωση την περιφερειακή των Αφρικανικών οικονομιών. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να υπάρξουν σοβαρές αλλαγές στις αφρικανικές οικονομίες, κάτι το οποίο σημαίνει στρατηγικό σχεδιασμό και περιφερειακή ολοκλήρωση. Και απαιτεί πάνω απ' όλα να υπάρχει μια συνεργασία των αφρικανικών κρατών για να επαναλάβουμε αυτό το οποίο έχει επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρώπη αλλά οι άλλες μεγάλες ε, προκλήσεις ε, που αφορούν τις προσπάθειες περιφερειακής ε, ανάπτυξης της Αφρικής αφορούν το εξής. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος αποτελείται από διάφορες περιφερειές και θα πρέπει να σεβόμαστε τους εμπορικούς μας εταίρους. Στην περίπτωση της Αφρικής αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι εμπορικές μας υποχρεώσεις να συμμορφωθούν όχι μόνο με τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι σε εταίρους όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να τηρούμε και τα παγκόσμια εμπορικά καθεστώτα του ΠΟΕ, του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι Αφρικανοί έχουν μεγάλες ε, φιλοδοξίες ε, ε, και βεβαίως θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι συμφωνίες στρατηγικής ε, εμπορικής ε, συνεργασίας, ε, παίρνοντα οπωσδήποτε στις λεπτομέρειες. Θα ήθελα λοιπόν να πω κυρίες και κύριοι ότι όσο δεν καταλήγουν αυτές οι συνομιλίες τόσο θα αποτυγχάνουν οι αναπτυξιακές προσπάθειες στην Αφρική. Άρα αυτό σημαίνει ότι οι εταίροι της Αφρικής θα πρέπει να είναι πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα ζητήματα τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη μεταφορά τεχνολογίας, την πρόσβαση στις αγορές, ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων και διπλωμάτων έβρεσης τεχνίας. Τώρα, περνάμε στις ευκαιρίες για τον 21ο αιώνα. Ήδη λοιπόν στα πλαίσια του 21ου αιώνα η Αφρική βρίσκεται στα, στην απαρχή μιας νέας εποχής. Προσπαθούμε τώρα να προωθήσουμε περισσότερο την επιστήμη και την έρευνα όλο και περισσότερο στην Αφρικανική Ήπειρο βλέπουμε ότι η τεχνολογία εχμής προωθείται. Έχουμε νέους καινοτόμους τομείς, οι οποίοι αναδύονται όλο και περισσότερο και μία υπόσχεση όλων και περισσότερων επενδύσεων και όλο και πιο αποδοτικών επενδύσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να προσελκύσουμε παγκοσμίους επενδυτέ, Αυτό ήδη έχει γίνει. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη νέα αυτή εποχή που ξημερώνει για την Αφρική. Η Αφρική και οι Αφρικανοί ενώ τον 20ο αιώνα ήταν πάρα πολύ συχνά θύματα και υφίσταντο διάφορες καταστάσεις. Τον 21ο αιώνα όμως η Αφρική θα είναι πλέον στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας, της γνώσης με έμπορους και πολίτες οι οποίοι θα θέλουν να συνάψουν όλο και περισσότερες εταιρικές σχέσεις. Είμαι πεπισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργαστεί όλο και περισσότερο ως στρατηγικός εταίρος με την Αφρική. Προσβλέπω λοιπόν σε μια νέα εποχή πολύ έντονων εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο επίρων μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστούμε κύριε Γερουσιαστά για τις παρατηρήσεις σας. Ας περάσουμε τώρα στον εξοχότο κύριο Κνόντο Ντάνκ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Έχετε 10 λεπτά για να κάνετε την αρχική σας παρέμβαση και έπειτα θα ακούσουμε και τον τρίτο ομιλητή μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της Αφρικής κατά τον 21ο αιώνα. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τη διοργάνωση της σημερινής συνεδρίασης, μολονότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα απολογισμό των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής, γιατί αυτό πιστεύω ότι θα μας επέτρεπε πραγματικά να δούμε πώς θέλουμε να διαμορφώσουμε τις μελλοντικέ μας σχέσεις σε ένα κόσμο που μεταβάλλεται συνεχώς. Ακριβώς στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει τόσο η Αφρική όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δούνε πώς θέλουν να διαμορφώσουν τις μελλοντικέ σας σχέσεις. Όπως και στην Ευρώπη, έτσι και στην Αφρική θα έχουμε πολύ σημαντικές αλλαγές στον 21ο αιώνα. Δημογραφικές καταρχάς αλλαγές. Το ΜΕΝ μας λένε ότι η Αφρική θα γίνει η με τους περισσότερους πολίτες μέχρι το 2050. Η Αφρική λοιπόν θα αντιστοιχεί πάνω από το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και η Ευρώπη την ίδια περίοδο θα έχει έναν λόγο ένα προς 20 όσον αφορά τον παγκόσμιο πληθυσμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Αφρική όλο και περισσότερο θα γνωρίσει όλο και περισσότερους πολίτες. Επίση, πολύ σημαντικό ήταν ο αριθμό των νέων στην Αφρικανική Ήπειρο, πολύ μεγαλύτερος από ό,τι σε άλλες υπήρους. Ξέρετε ότι αυτό αποτελεί πολύ σημαντική πρόκληση, αλλά και σημαντική ευκαιρία. Πρόκληση γιατί θα πρέπει να δημιουργηθούν θέσει απασχόλησης, αλλά και ευκαιρία γιατί οι νέοι αυτοί θα καταφέρουν να προωθήσουν περισσότερο την καινοτομία. Η Αφρική στο παρελθόν ήταν κατά τη διάρκεια τη δεκαετία του 1960 κυρίω μια αγροτική οικονομία. Την εποχή εκείνη ανακτούσαν την ανεξαρτησία του σε περισσότερε αφρικανικέ χώρε. Στο μέλλον η οικονομία τη Αφρική ήταν όλο και περισσότερο αστική. Σύμφωνα με, το, με στοιχεία πάλι των Ηνωμένων Εθνών, ε, μέχρι το 2017 ήταν μικρότερος αριθμός των ε, Αφρικανών οι οποίοι ζούσαν σε πόλεις σε σχέση με τον αριθμό των Ευρωπαίων. Αλλά η τάση αυτή θα αντιστραφεί. Χρειάστηκε 110 χρόνια προκειμένου η Ευρώπη να καταφέρει να φτάσει ένα ποσοστό του 40% όσον αφορά τον αστικό της πληθυσμό. Σε ένα μισό αιώνα, σε 50 χρόνια, έγινε η σημαντική αυτή αλλαγή στην Αφρικανική Ήπειρο. Γνωρίσαμε λοιπόν μία ραγδαία αστικοποίηση του πληθυσμού μα, των κοινωνιών μα, πράγμα το οποίο θέτει τεράστιε προκλήσει όσον αφορά την οργάνωση τη οικονομία μα, όσον αφορά τα εκπαιδευτικά μα συστήματα, όσον αφορά τα συστήματα απασχόληση. Έχουμε πόλει οι οποίε αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα και υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στην μεγέθυνση των πόλεων και τι αντίστοιχε κρατικέ υπηρεσίε. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πάρα πολλέ άτυπε ζώνε ε, κατοικιών οι οποίες δεν, δεν διέπονται από αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης ακόμα. Το δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να θίξω είναι η οικονομία. Η αφρικανική οικονομία βασίζεται προφανώς και εξαρτάται από την παγκόσμια οικονομία. Ο τεράστιος πλούτος της Υπήρους μου μέχρι σήμερα δεν έχει τύχει πλήρους εκμετάλλευσης. Και όταν εκμεταλλευόμαστε τον πλούτο αυτό, αυτό γίνεται με έναν τρόπο ο οποίο είναι ιδιαίτερα βάναυσος και ο οποίος τελικά δεν επιφέρει πλούτο στην ίδια την Αφρικανική Ήπειρο. Γι' αυτό το λόγο ένα μεγάλο τμήμα του αφρικανικού πληθυσμού ζει στα όρια τη φτώχεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν στο Μόλο να υπάρχει μια απαραίτητη τεχνολογική μεταφορά προκειμένου να μετασχηματίσουμε την αφρικανική οικονομία, να την αξιοποιήσουμε επί τόπου, να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία και να επιλύσουμε το ακαθόδε πρόβλημα τη απασχόληση πρόβλημα το οποίο δημιουργείται τέτοια τεράστια έξοδο από τις ε, αγροτικές περιοχές προς τα αστικά κέντρα ή ολότελα από την Αφρική προς την Ευρώπη. Τρίτη σημαντική ε, πρόκληση, κοινωνικοπολιτική. Κάθε φορά που μιλάμε για την Αφρική θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί μιλάμε για μια Ήπειρο, όπου οι ανεξάρτητες χώρες υφίστανται περίπου εδώ και 50 χρόνια. Από την άποψη λοιπόν αυτή, η Αφρική βρίσκεται ακόμα σε φάση θεσμικής εξέλιξης και διαμόρφωσης. Δεν μπορούμε λοιπόν να αναλύουμε την Αφρική με τον ίδιο τρόπο και τα ίδια μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε για παλαιότερες χώρες, για τις οποίες είχαμε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θεσμικής ορίμανσης. Πολλές φορές υπερβαίνει 100 χρόνια. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Αφρική. Μετά από αρχική, μια, μια αρχική περίοδο 20 ετών, που χαρακτηρίστηκε κυρίως από, μια πολύ σημαντική, από ένα πολύ σημαντικό κεντρικό χαρακτήρα της εξουσίας, περνάμε σε μια νέα εποχή που χαρακτηρίζεται περισσότερο από την προσχώρηση των κρατών της Αφρικής σε πιο πλουραλιστικά πολιτικά συστήματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε πολιτικό επίπεδο ακολουθούμε όλο και περισσότερο δημοκρατικά συστήματα, ότι πρέπει να γνωρίσουμε αυτό. Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε πολιτικές κρίσεις σημαντικές σε διάφορες χώρες Αφρικής. Η αποκέντρωση πάντως της εξουσίας λαμβάνει χώρα στις περισσότερες χώρες και ενισχύει όλο και περισσότερο το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, το οποίο μπορεί να έχει στρατηγική συμβολή στην εκχώρηση εξουσιών προς, από το κέντρο προς τις ε, τοπικές ε, περιφερειακές αρχές. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την εξέλιξη της οικονομίας και την εξέλιξη της κοινωνίας. Το κράτος δικαίου ενισχύεται όλο και περισσότερο. Αντιμετωπίσουμε παρόλα αυτά κοινωνικοπολιτικές δυσκολίες που απορρέουν από το ότι τα κράτη δεν είναι σε θέση να τηρήσουν τι δεσμεύσει του όσον αφορά τον εξυγχρονισμό των κοινωνιών, βασική υπόσχεση που είχε δεθεί πριν από πολλά χρόνια σε διάφορες χώρες Αφρικής. Δεν ακολουθήθηκαν όμως οι απαραίτητες δημόσιες πολιτικές, οι οποίες δώσανε πολύ μεγαλύτερη σημασία τελικά στην ικανοποίηση των αναγκών και των επιτάξεων της οικονομίας και του κεφαλαίου και, όχι, και δεν αποκρίθηκαν τόσο πολύ στις ανάγκες της κοινωνίας. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν ε, τεράστιες θύλακες στις κοινωνίες που τελικά νιώσανε ότι είχαν εγκαταλειφθεί εντελώς από την κεντρική εξουσία. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να οργανωθούμε λίγο περισσότερο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο στην Αφρική προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα δεινά της παγκοσμιοποίησης. Γι' αυτό το λόγο αρχίσαμε σιγά σιγά να προωθούμε μία διαδικασία περιφερειακής ολοκλήρωσης της Αφρικανικής Υπήρου προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον κατακαιρματισμό που είχαμε συναντήσει στο παρελθόν. Μέσω της οικονομικής αυτής περιφερειακής ολοκλήρωσης μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερο τις αρμονικές οικονομικές αλλαγές σε επίπεδο Αφρικανικής Υπήρου. Α μην ξεχνάμε ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στα πλαίσια της Αφρικανικής Υπήρου από το 1963 συναντώνται δύο φορές το χρόνο προκειμένου να συζητήσουν κοινά ζητήματα και κοινέ ανησυχίες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δίνει ιδιαίτερη νομιμότητα στην δράση της Αφρικανικής Ένωσης η οποία αντικατέστησε τον Οργανισμό Αφρικανικής Ένωσης. Το 2016 είδαμε ότι προσχώρησε στην Αφρικανική Ένωση και το Βασίλειο του Μαρόκου. Κατά αυτόν τον τρόπο πλέον όλα τα κράτη της Αφρικής συμμετέχουν στην Αφρικανική Ένωση και μπορούν κατά αυτόν τον τρόπο να συνδιαλέγονται μέσω της Αφρικανικής Ένωσης με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Θεωρώ λοιπόν ότι σε πολιτικό επίπεδο κινούμαστε σωστό δρόμο, μολονότι μπορούμε να έχουμε μεμονωμένες κρίσεις και μεμονωμένα προβλήματα. Ο Παναφρικανικό αυτό διάλογο που έχουμε θεσπίσει συμβάλλει πάρα πολύ στο να μειωθούν οι συγκρούσεις και να υπάρχει μια, ένα διάχυτο πνεύμα πλέον ειρήνευση στην Ήπειρο. Εμείς ονειρευόμαστε τη στιγμή εκείνη που βασιζόμενοι πλέον στις αμοιβέ εμπειρίες μας θα καταφέρουμε τελικά στα πλαίσια της Αφρικανικής Ένωσης να αντιμετωπίσουμε την Ήπειρό μας ως μια ενιαία Ήπειρο παρότι υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των χωρών μας. Ακριβώς με τον τρόπο που και εσείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μολονότι απαρτίζεστε από διαφορετικά κράτη-μέλη, λειτουργείτε ως μία κοινή ένωση. Έχουμε τέλος στα πλαίσια της Αφρικανικής Ένωσης και ένα κοινοβούλιο, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, όπου προσπαθούμε οι ε, βουλευτές από τις Αφρικανικές χώρες να μιλάμε με μία ενιαία φωνή και να εκπροσωπούμε σε διεθνή φόρα τους πολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάμε τώρα για να ακούσουμε τον τρίτο ομιλητή σήμερα στο πάνελ ο Περιφερειακός Διευθυντής ε, του Διεθνούς Οργανισμού για την ε, Μετανάστευση, ο κύριος Αμπρόζη, και εσείς έχετε 10 λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την δυνατότητα αυτή που μου δίνετε να είμαι εδώ σήμερα μαζί σας για να συζητήσουμε προκλήσεις και ευκαιρίες που εμφανίζονται στις σχέσεις μας με την Αφρική και για την ίδια την Αφρική καθότι προσεγγίζουμε και το, τη σύνοδο στο Αμπιτζάν και είναι μια κατάλληλη χρονική στιγμή να δούμε πού βρισκόμαστε, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ποιες είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που μπορεί να έχουμε για το μέλλον. Αυτό θα το κάνω βέβαια υπό την έννοια της κινητικότητας και της μετανάστευσης που είναι η δική μας συνεισφορά προς τη ζήτηση αυτή και να ξεκινήσω με ένα πλαίσιο. Οι περισσότερες πληροφορίες ήδη αναφέρθηκαν από τους άλλους ομιλητές. Η Αφρικανική Ένωση είναι η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη ήπειρος σήμερα με περί το 16% του παγκόσμιου πληθυσμού και επίσης είναι μια Ήπειρος που είναι από τις νεαρότερες ως προς τον πληθυσμό και με έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους δείκτες πληθυσμού σε σχέση με τις άλλες ήπειρους Στην Ευρώπη έχουμε ακριβώς το αντίστροφο. Μία από τις παλαιότερες πληθυσμιακά υπήρους και που λιγότερο αυξάνει τον πληθυσμό της. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί στα πλαίσια της συζήτησης της κινητικότητας και μετανάστευσης πολύ συχνά ακολουθούμε κάποιες έτσι υπεραπλουστευτικές προσεγγίσεις και ενδεχομένως να μην είμαστε απόλυτα ακριβείς ή απόλυτα υπεύθυνοι οδηγώντας σε μια σειρά από αρνητικές αντιδράσεις επί τη βάση αξιολόγησης της πραγματικότητας που δεν συμπίπτει απολύτως με την αλήθεια. Αν δούμε τα τελευταία χρόνια θα συνειδητοποιήσουμε ότι η μετανάστευση δεν έχει αυξηθεί από την Αφρική τόσο δραματικά όσο ακούμε, ίσως πρόσφατα και αν δούμε αυτό που περιγράφεται ως βασικότερο πρόβλημα μετανάστευση για την Ευρώπη, ακούμε για χιλιάδες Αφρικανούς που είναι έτοιμοι να διασχίσουν τη Μεσόγειο και να φτάσουν στην Ευρώπη, ακούμε λέξεις όπως εισβολή, όλα αυτά δίνουν την εντύπωση μιας έτσι άμυνας, ενός κλεισίματος. Κατά μεγάλη πλειοψηφία να πω ότι οι Αφρικανοί καταρχάς μετακινούνται εντός της Αφρικανικής Υπήρου. Επίσης είναι σημαντικό να διαφοροποιήσουμε τις τάσεις της μετανάστευσης ανάλογα με την περιοχή της Αφρικής η αχάριος κινείται προς το βορρά, η Βόρεια Αφρική έχει πολύ διαφοροποιημένες κινήσεις και προς την Ευρώπη, αλλά και προς τις χώρες του κόλπου, προς την Αμερική και προς την Ασία σε σημαντικό μάλιστα βαθμό. Και μαζί με τις διάφορες τάσεις υπάρχουν διάφορες ομαδοποιήσεις κινήσεων, άνθρωποι που αναζητούν άσυλο άνθρωποι που προσπαθούν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση, που θέλουν να επανανοθούν με την οικογένειά τους, που είναι θύματα λαθρεμπορίας ανθρώπων, που είναι από τις βασικές μάστιγες της εποχής. Υπάρχουν, εν περιπτώσει, διάφοροι λόγοι που οθούν τους ανθρώπους να μετακινούνται. Σημαντική όμως πτυχή Ω προ το γενικότερο πλαίσιο είναι ότι η Αφρική σήμερα είναι η Ήπειρος που φιλοξενεί το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων και εσωτερικά μετακινωμένων για διάφορους λόγους. Συζητώντας λοιπόν στο πλαίσιο αυτό, καλό είναι να λαμβάνουμε υπόψη μας την πραγματικότητα και να μην δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα διάφορα μυθεύματα ή πλαστές εικόνες που μεταδίδονται, ιδιαίτερα όταν λαμβάνουμε αποφάσεις πολιτικής σχετικά με την Αφρική και με διάφορα άλλα μέρη του κόσμου. Επομένως, πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι πρέπει να καταβάλουμε μια σημαντική προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις μας θα λαμβάνονται επί τη βάση αποδείξεων και όχι κάποιας Εντύπωση με κάποιο βραχυπρόθεσμο ή άλλο πολιτικό όφελος. Τώρα βλέπω ότι έχω χάσει το μισό μου χρόνο, οπότε ας επιταχύνω. Το όφελος που βλέπουμε στην σωστή διαχείριση της κινητικότητας και της μετανάστευσης και κάποιες ε, γρήγορες συστάσεις. Η Ευρώπη γνωρίζει πολύ καλά από την δική της ιστορία ότι η μετανάστευση είναι μια πολιτική μετρίασης της ένδυας, αντιστάθμισης της πίεσης επί του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος μιας χώρας, υπό κάποιες έννοιες μια στρατηγική επιβίωσης. Αυτό το ξέρει καλά η Ευρώπη, διότι αυτό ακριβώ έκανε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με μεγάλης κλίμακας μετανάστευση προς πρώτα απ' όλα την Αμερική, και τη Βόρεια αλλά και την Νότια και επομένως και εμείς οι ίδιοι πριν από μία γενιά και ούτε χρησιμοποίησαμε την ίδια στρατηγική για να απαλύνουμε την πίεση που δεχόμασταν στις κοινωνικές και οικονομικές μας δομές. Η αντιστάθμιση λοιπόν της πίεσης και η δημιουργία ευκαιριών κοινωνικών και οικονομικών για τους μετανάστες αλλά και για τις χώρες και προέλευσης και προορισμού των μεταναστών αυτών. Ιδιαίτερα σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντική μείωση εν πάση αλλαγή πορείας της δημογραφικής καμπύλης όπου επίσης εντοπίζουμε σημαντικά κενά στην αγορά εργασίας ζητούμε εργατικό δυναμικό που δεν είναι διαθέσιμο, που δεν είναι παρόν στην Ευρώπη, επομένως για την ίδια μας την οικονομική μεγέθυνση πρέπει να δούμε τη μετανάστευση και τη διαχείρισή της σε υποδιαφορετικό φως. Τώρα, όσον αφορά την αντιστάθμιση της ένδυας για τα νοικοκυριά και της κοινωνίας για τους ίδιους τους Αφρικανούς, τα εμβάσματα που αποστέλουν στα σπίτια τους στις ε, κοινότητές τους είναι πολύ υψηλότερου όγκου από τους διάφορους οργανισμούς αναπτυξιακής βοήθειας που ενεργοποιούνται στις χώρες αυτές. Είναι λοιπόν σημαντικό να αξιοποιούμε τις πολιτικές μας σε σχέση με το όφελος που οι αφρικανικές χώρες και οι Αφρικανοί δέχονται ως βοήθεια από τους πολίτες τους που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Ο τρόπος λοιπόν τον οποίο λειτουργεί η διασπορά γενικώ είναι θεμελιώδης σημασία για την ανάπτυξη συγκεκριμένων κοινωνιών στην Αφρικανική Ήπειρο. Τώρα, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευση και ιδιαίτερα μετανάστευση από την Αφρική, πρέπει να πούμε ότι πρώτα απ' όλα όλα τα κράτη έχουν αναλάβει πολλαπλές δεσμεύσει σε διεθνές επίπεδο με, το, με, με τους στόχους SDG καταρχά, όπου οι όγκοι της μετανάστευση είναι σε υψηλό σημείο ιεράρχησης τη μεγιστοποίηση τη αναπτυξιακής βοήθεια που ελήφθη ω δεσμευσή από το Σύνδεσμο Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρυσι πάλι στη Νέα Υόρκη με την ε, διακήρυξη τη Νέα Υόρκης η διεθνή κοινότητα μαζί με όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράμμισαν μια σειρά από αρχέ και αξίε για τη μεγιστοποίηση των, του ωφέλους της μετανάστευσης. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά που κάνουμε θα είναι συνεπές προς τις δεσμεύσεις αυτές που έχουμε αναλάβει. Δηλαδή, όταν λαμβάνουμε μια απόφαση για την εσωτερική διάσταση της μετανάστευσης στην Ευρώπη, αυτές οι αποφάσεις δεν θα πρέπει να αντιφάσκουν προς δεσμές που έχουμε λάβει για την εξωτερική διάσταση και δεν θα πρέπει να, είναι, να στρέφονται εναντίον του συμφέροντος των Αφρικανικών χωρών μαζί με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει στην σύσταση εταιρικών σχέσεων που σημαίνει ισότιμη σχέση, που σημαίνει ότι τα συμφέροντα λαμβάνονται υπόψη στο ίδιο επίπεδο με ισότιμο και δίκαιο τρόπο και χωρίς να χρησιμοποιούνται ως μόχλευση ώστε να επιτευχθεί κάποιο πλεονέκτημα εις βάρος της άλλης πλευράς. Νομίζω ότι η συνέπεια της πολιτικής για τη διαχείριση της μετανάστευσης και της εταιρικής σχέσης με την Αφρική για θέματα μετανάστευσης είναι ουσιώδους σημασία. Υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν στο πλαίσιο αυτό και είμαι πεπισμένο, λέει ο μιλητή, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ηγηθεί του δρόμου προς την καλύτερη υλοποίηση των μέσων που έχει διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να δημιουργήσει μια πολύ πιο ισχυρή εταιρική σχέση με την Αφρική επί τη βάση της ισότητος και των πραγματικά κοινών στόχων και οραμάτων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τους τρεις ομιλητές μας. Ας ακούσουμε τώρα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Γκάλερ θα πάρει πρώτος το λόγο, ο οποίος δεν είναι απλώς μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Άρα γνωρίζεστε πολύ καλά, έτσι δεν είναι. Κύριε Γκάλερ, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Yeah, um, attention, je vais parler en allemand. <laughs> Um, Κύριε, μιλήσω γερμανικά. Zunächst in meiner Funktion als Vorsitzender Πρώτα απ' όλα ως ε, πρόεδρος ε, της αντιπροσωπείας για σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο θα ήθελα να καλωσορίσω τους συναδέλφους ε, ε, και στον πρόεδρο του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Ροζέ Γκόντο Ντάν. Και χαίρομαι που έχετε έρθει και έχουμε μεγάλες αντιπροσωπείες από το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, αλλά και συναδέλφους από την Ιγυρία, το Μαρόκο, την, την Ισία. Θεωρώ ότι αυτό αναδεικνύει το ενδιαφέρον για διάλογο, αλλά από την άλλη ότι και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνουμε ότι οι σχέσεις ε, με την Αφρική είναι σημαντικές. Επίσης, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον κύριο Ταγιάννη, για την πρωτοβουλία του αυτή και πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς. Το να στρέψουμε την προσοχή μας στην Αφρική είναι δύσκολο για την Ευρώπη. Υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται και αναδεικνύουν τη σημασία των σχέσεων, αλλά δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην ευρύτερη κοινωνία. Πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον προς Νότον. Είναι σημαντικός γείτονας η Αφρική και η μοίρα μας συνδέεται στενά με την Αφρική και πρέπει να διευρύνουμε το βλέμμα μας πέρα από τα επίκαιρα προβλήματα. Πολλοί Ευρωπαίοι όταν ακούν Αφρική σκέφτονται μια κρίση προσφυγική, αλλά βεβαίως αυτό είναι τελείω ε, κοντόφθαλμο. Έχουμε ένα ευρύτατο πεδίο κοινή ευθύνη. Γι' αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία εδώ να έχουμε κάποιες ανταλλαγές απόψεων με τους συναδελφούς. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε μια συνάντηση με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο στο Αμπιτζάν και αυτό νομίζω είναι μια έκφραση της σημασίας ε, που αποδίδουμε. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα την προ-σύνοδο κορυφής ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής και Αφρικανικής Ένωσης και θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για αυτήν την καλή συνεργασία και για το ότι αφαιρνόμαστε στα θέματα που είναι σημαντικά και το θέμα της επένδυσης στην νεολαία που βεβαίως θα κυριαρχήσει στην Αμπιτζάν είναι ένα θέμα που αφορά και όλα τα υπόλοιπα θέματα γιατί η νεολαία έχει το μέλλον μπροστά της και για την νεολαία και με την νεολαία πρέπει να δούμε αυτά τα ζητήματα. Είχαμε την ε, προπροηγούμενη εβδομάδα εδώ μια διάσκεψη των οργανώσεων της νεολαίας από Αφρική και Ευρώπη και είχαμε κάνει πολλή δουλειά για το θέμα αυτό ε, γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το τι θέλει και η νεολαία από τους πολιτικούς στο Αμπιτζάν και ελπίζω και εύχομαι να τα βλέπουμε αυτά όχι μόνο εν ώψη της ε, Συνόδου Κορυφής αλλά και μετά παραπέρα ως βουλευτές ε, να πιέσουμε την εκτελεστική εξουσία να μην κάνει μόνο δηλώσεις της Συνόδους Κορυφής, αλλά να εφαρμόζει και όλες ε, τα συμφωνημένα. Αυτό είναι προς το κοινό συμφέρον μας και αυτή είναι η δουλειά μας ως βουλευτές και γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω τη στήριξή μου στους συναδέλφους από την Αφρική και όπως είπα πρέπει να συνεχίσουμε να φέρνουμε αυτό το θέμα στο προσκήνιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και βεβαίως αναμένω την περαιτέρω συζήτηση και αυτήν και την επόμενη εβδομάδα. Περνάμε στον κύριο Παντσερή από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκπροσωπώντας την Προεδρία της Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είμαι και εγώ πεπισμένος ότι οι σχέσεις με την Αφρική είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ωστόσο υπάρχουν κάποια μηνύματα που προέρχονται από την Αφρική, από την Κένια, την Λιβερία, μέχρι και την Ζιμπάμπουε που μας δείχνουν μια Ήπειρο που προσπαθεί να βρει το μέλλον της δημοκρατικός αλλά εκτός των γνωστών μονοπατιών και δεν τα καταφέρνει. Διάφορα κρούσματα μεταξύ των οποίων της Χαράρε δείχνουν πόσο δυνατή είναι, πόσο δυνατή είναι μια τάση έτσι, στρατιωτικών πραξικοπημάτων και δεσποτισμού γενικά. Επομένως, ο νέος δρόμος, ο δρόμος προς την δημοκρατία θα πρέπει να στηριχθεί και από τα εθνικά κοινοβούλια με όλη την προσπάθεια που αυτό απαιτείται. Και επομένως θα ήταν πολύ χρήσιμο πιστεύω να ακούσουμε τη δική σας άποψη στη δημοκρατική μεταξέλιξη που πρέπει μπορεί και πρέπει να έχει η Αφρικανική Ήπειρος. Τώρα, οι συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών υπήρξαν, όπως είπαν πολλοί ομιλητές, πολύ σημαντικός μοχλός για να ενισχύσουμε την συνεργασία μας και την ανάπτυξη. Αλλά μιλώντας για ανάπτυξη, εγώ δεν θα ήθελα να εννοώ μόνο το επιχειρήν, την business, αλλά και την ανθρώπινη διάσταση. Και νομίζω ότι όλο και πιο δύσκολα μπορεί κανείς να αποδεχθεί κάποιες ερεσιμότητες που τίθενται στο περιθώριο των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών και πιστεύω ότι θα ήταν πολύ κατάλληλο αυτό το σημείο προς συζήτηση αυτή την εβδομάδα που βρίσκεστε εδώ. Ο αντίκτυπος επί του πληθυσμού των πολιτών διαφόρων από τις συμφωνίες αυτές ελευθέρων συναλλαγών είναι και αυτά ή στο πλαίσιο της εξέτασής μας της κινητικότητας. Πολύ συχνά πλήττουν οι πολιτικές μετανάστες ε, της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αλήθεια ότι θα φανεί τελικώς πόσο ανάγκη έχουμε την μετανάστευση. Και είναι σημαντικό να μιλούμε για τη δημογραφική εξέλιξη της Αφρικής, όχι για να ξέρουμε πόσοι άνθρωποι μπορεί να έρθουν εδώ, αλλά για να ξέρουμε πώς μπορούμε με καλύτερο τρόπο να χειριστούμε το επίπεδο διαβίωσης, αξιοπρεπούς διαβίωσης για, τις, ε, για τους πολίτες, τους κατοίκους της Υπήρου αυτής και των χωρών αυτών και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα αρνητικά Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση των διμερών επαφών και σχέσεών μας που να βάζουν στο κέντρο της συζήτησης αυτά τα θέματα. to... Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Καστάλντο από το EFDD παρακαλώ. Σας ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω τους ε, προσκεκλημένους μας ε, από το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο αλλά και από άλλα Αφρικανικά Κοινοβούλια είδα ότι έχει και μια αντιπροσωπεία εδώ πέρα από την Τινησία και την Ιγυρία. Και πολλές φορές ως Ευρωβουλευτής έχω πάει στις χώρες αυτές στα πλαίσια αποστολών. Ιστορική στιγμή λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις σχέσεις της με την Αφρική. Δέκα χρόνια πέρασαν από την έγκριση της κοινή στρατηγικής Αφρικανικής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο αυτές ενώσεις μας στις 23 Νοεμβρίου θα έχουν την πέμπτη τους πλέον σύνοδο. Τα ακόλουθα ερωτήματα θα ήθελα να θέσω προς τους καλεσμένους μας. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται στο μέλλον η μεταξύ μόν σχέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την άποψή σας διαμορφώνει σωστά τη σχέση με την Αφρική. Πώς θα πρέπει να επαναπροσαρμοστεί η στρατηγική αν πιστεύετε ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί. Και αν θεωρείτε ότι ε, δεν ακολουθούν το σωστό δρόμο οι πολιτικές μας. Όπως υπόθηκε και πριν από λίγο, θα ήθελα και εγώ να το τονίσω αυτό μέσω του ερωτήματός μου. Δίδεται η γενικότερη εντύπωση ότι αυτό το σχέδιο Marshall για την Αφρική, το οποίο αναφέραμε και συζητήσαμε πριν πολλά χρόνια εδώ στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, η λεγόμενη εξωτερική επένδυση, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα μέσα. Πιστεύετε πραγματικά λοιπόν ότι το σχέδιο αυτό Marshall και τα επενδυτικά αυτά μέσα λειτουργήσαν τελικά μόνο βραχυπρόθεσμα με απότερο στόχο να κρατήσουν τους μετανάστες στην Αφρικανική Ήπειρο χωρίς να συμβάλλουν πραγματικά στη μακροπρόθεσμη πύληση των προβλημάτων της Ήπειρου. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα, τα μέσα αναπτυξιακής βοήθειας και όσον αφορά έπειτα την νεολαία, κάτι το οποίο θίξτε πριν από λίγο. Η νεολαία είπατε ότι θα είναι ένα από τα σημαντικότερα επόμενα ζητήματα που θα έχουμε στην επερχόμενη Σύνοδο Αφρικανικής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμουνα και εγώ στην Αμπιτζάν πριν από μερικές εβδομάδες για την προπαρασκευαστική αυτή συνεδρίαση για τη νεολαία. Και είμαι πεπισμένο όταν μιλάμε για νεολαία, μιλάμε ουσιαστικά για τους ανθρώπους που θα κληθούν στο μέλλον να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως η ε, ριζοσπαστικοποίηση, η τρομοκρατία. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να εμπλέξουν περισσότερο και τους νέους και τις τοπικές κοινότητες στα ζητήματα αυτά. Ξέρουμε παράλληλα ότι η εκπαίδευση και η ανάπτυξη είναι η καλύτερη θεραπεία για την αντιμετώπιση της ε, τρομοκρατίας. Ως προς αυτό, πώς πιστεύετε ότι έχει ε, εμπλέξει η συνεργασία της Αφρικανικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους νέους. Τι πιστεύετε όσον αφορά την ενσωμάτωση των νέων περισσότερο στη μεταξύ μόνο συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις, γιατί νομίζω ότι οτιδήποτε επινοούμε σε θεωρητικό επίπεδο θα πρέπει να αντιστοιχεί τελικά σε μια έμπρακτη εφαρμογή. Νομίζω ότι δεν μπορούμε εμείς να επινοούμε και να καταρτίζουμε σχέδια συνεργασίας χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη πραγματικά αυτά τα οποία έχουν να πούν οι πληθυσμοί μας και από τις δύο πλευρές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας και ελπίζω ότι ε, η μεταξύ ημών συνεργασία πραγματικά θα αντικατοπτρίζει και θα καθρεφτίζει τη φιλοδοξία της Ευρω... Ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης για την μετεξέλιξη των σχέσεών τους. Σας ευχαριστούμε κύριε Καστάλντο. Μπορούμε τώρα να ακούσουμε και άλλους ευρωβουλευτές εφόσον θέλουν να πάρουν το λόγο ή καλεσμένους μας και από το Μαρόκο, την Τινησία ή την Ιγυρία. Ζητώ συγγνώμη, δεν γνωρίζω το όνομά σας, αλλά αν σηκώσετε το χέρι θα σας δώσω το λόγο. Ο κύριος στο βάθος, παρακαλώ. You just have to press the button to have the micro come on. Yeah. Είστε απλώς το κουμπί για να ενεργοποιηθεί το μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε σαν τα από το Κοινοβούλιο της Νιγηρίας. Πήρα το λόγο για να μιλήσω για το πρόβλημα της μετανάστευσης. Έχουμε πάρα πολλά φόρα στα οποία συζητάμε το πρόβλημα της μετανάστευσης κυρίως ε, από την Αφρική προς άλλες χώρες. Δυστυχώς υφίστανται ακόμα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν ε, και τα οποία ουσιαστικά δεν, με τα οποία δεν ασχολείται ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με τα ζητήματα αυτά. Στην Αφρική έχουμε τέσσερις χώρες, τέσσερις περιοχές που από στρατηγικής πλευράς είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Νιγηρία, Δυτική Αφρική, Νότιος Αφρική, Ανατολική Αφρική, Αίγυπτος, τη Βόρεια Αφρική και Αιθιοπία στο κέρας Αφρικής. Οι τέσσερις αυτές χώρες που εντάσσονται στις τέσσερις αυτές περιοχές Αφρικανικής Επίρου είναι περιοχές με τις οποίες θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει σε αυτές να δημιουργηθούν οι κατάλληλες στρατηγικές υποδομές και επαφιόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να ασκήσει πίεση για το ζήτημα αυτό. Αν υπήρχαν οι απαραίτητε στρατηγικέ υποδομέ στι τέσσερι αυτέ χώρε και κατ' επέκταση στι τέσσερι αυτέ ευρύτερε γεωγραφικέ περιοχέ, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών θα μπορούσαν ε, εύκολα να βρουν μια θέση απασχόληση και να κερδίσουν τα προστοζήν στι ίδιε τι χώρε του. Θα μπορούσε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προσπαθήσει να εξορροπήσει λίγο την οικονομία των χωρών της Νοτιού Αφρικής με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής αυτής να μην έχουν κανένα λόγο πλέον να εγκαταλείψουν την περιοχή τους και να ψάξουν τελικά Θέσει απασχόληση σε άλλες χώρες ή σε άλλες περιοχές. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και με τη δική μου τη χώρα, με την Ιγυρία. Ξέρετε ότι αν υπήρχαν οι απαραίτητε επενδύσεις και απαραίτητε υποδομές θα μπορούσαμε να είχαμε έναν τόσο αναπτυγμένο βιομηχανικό τομέα που θα μπορούσε πραγματικά να παρήχε επαρκή θέση απασχόληση για όλο τον ενεργό πληθυσμό. Το ίδιο ισχύει και για την Αίγυπτο. Μια χώρα που αντιμετωπίζει σημαντικότερε προκλήσει ασφάλεια. Και έχουμε έπειτα και την Δυτική Αφρική και την γενικότερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούσε να επέμβει τρόπον την ώστε να εγγυηθεί τη σταθερότητα των περιοχών αυτών, δεν θα φεύγανε τόσοι πολλοί κάτοικοι από αυτές τις περιοχές ε, για να έρθουν εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα την πρόκληση της έμβια, την αντιμετώπιση της φτώχειας, ε, αν δεν βελτιωθεί η οικονομία στην Ήπειρό μας, ε, και δεν καταφέρουμε να έχουμε την απαραίτητη απασχόληση στην Αφρικανική Ήπειρο, χώρες όπως η Σομαλία και άλλες χώρες δεν πρόκειται να καταφέρουν να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Με την απαραίτητη οικονομική ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές δεν πρόκειται να υπάρχει τόσο έντονη μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο θα πρέπει να επέμβει να ασχοληθεί με τα ζητήματα αυτά, να κρούσει τον κόδωνα κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει τις επικοδομητικές αυτές παρεμβάσεις στην Αφρική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Γερουσιαστά. Πρωτού δώσω το λόγο ε, στα μέλη του πάνελ ε, να προσθέσω και ένα-δύο δικά μου ερωτήματα. Καταρχάς για τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε εμπορικές πολιτικές, πολιτικές αλληλείας, υδατοκαλλιέργειας κτλ. Και έχω την εντύπωση ότι κάποιες φορές αυτές οι πολιτικές παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη σε κάποιες από τις χώρες σας. Κατά πόσον δηλαδή η πολιτική μας αλληλείας μεταξύ άλλων είναι υπερβολικά επιθετική για κάποιες παράκτιες περιοχές της Αφρικής. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε για να αντισταθμίσουμε την οικονομική μεγέθυνση που χρειάζεται και ο νέος πληθυσμός σας. Και άλλη μια ερώτηση, προτού δώσω το λόγο, είναι ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία. Μιλώ ως ευτυχής σύζυγος, αλλά πολλές φορές ακούμε ότι μάλλον είναι από τα στοιχεία που θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε από κοινού, νομίζω. Τώρα σας ευχαριστώ που ακούσατε και τις δικέ μου ερωτήσει. Ας πάμε αντίστροφα, οπότε ξεκινάω από εσά αν δεν έχετε αντίρρηση. Ε, σας ευχαριστώ. Κάποια γρήγορα σχόλια στα όσα ελέγχθησαν. Πρώτα απ' όλα, σχετικά με το γεγονός ότι η πλειοψηφία των Αφρικανών μεταναστών βρίσκεται ακριβώς στην Αφρική και όχι στην Ευρώπη. Και ακριβώ ε, επ' αυτού τοποθετήθηκε και το αξιότιμο μέλο ε, του Κοινοβουλίου. Αυτό προσπαθούσα να πω ε, λέγοντα ότι η εταιρική σχέση μεταξύ Αφρική και Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι μια πραγματική, ισότιμη εταιρική σχέση. Υπάρχει υπερβολική ανησυχία, εκφράζεται υπερβολική ανησυχία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη να αμυνθούμε ε, έναντι κάποιου κινδύνου της έλευσης δηλαδή των μεταναστών και ξεχνούμε κάποιες άλλες υποχρεώσεις που είναι πιο σημαντικές, μία από τις είναι να συνεργαστούμε με τις αφρικανικές χώρες ώστε να διαχειριστούμε ακριβώς το θέμα της κινητικότητας που έχουν στις χώρες τους. Και τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αρκετές περιπτώσεις βλέπουμε καθημερινά τι συμβαίνει στους μετανάστες στη Λιβύη. όπου πολλούνται σε σύγχρονα σκλαβοπάζαρα. Και είναι κοινή ευθύνη, νομίζω, των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τη, των όλων των Εθνικών Κοινοβουλίων μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, να προστατεύσουν τους ανθρώπους αυτούς που έχουν γίνει θύματα και νομίζω ότι αυτό το στοιχείο δεν είναι όσο παρόν θα έπρεπε να είναι στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να φύγουμε λιγάκι από την αιμονή με τους αριθμούς, πόσοι φεύγουν, πόσοι έρχονται κτλ. Και να κάνουμε προτεραιότητά μας τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών, των προσφύγων και των ίδιων των πολιτών μας για το μέλλον βεβαίως ε, τις σχέσεις με την Αφρικανική Ένωση θα δώσω το λόγο σε πολύ αρμοδιότερους από μένα, αλλά για τα θέματα της μετανάστευσης πιστεύω ότι αυτό είναι από τα σημαντικότερα σημεία. Αν είναι να έχουμε μια πραγματικά κοινή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, θα πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι συνδίκες διαβίωσης των πολιτών μας, όλων των πολιτών μας, να είναι στο επίκεντρο. Μία άλλη στρεβλωμένη αντίληψη που υπερισχύει είναι ότι η οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να σταματήσει τη μετανάστευση. Δεν ισχύει. Ε, το έχουμε δει πολλαπλές φορές σε όλο τον κόσμο και το αποδεικνύουμε εμείς εδώ. Εγώ ε, είμαι εκτός της χώρας μου τα τελευταία 29 χρόνια η οικονομική ανάπτυξη δεν σταματάει και δεν θα έπρεπε. Δεν υπάρχει ένας λόγος γιατί να σταματάει τη μετανάστευση. Οι άνθρωποι μετακινούνται και θα έπρεπε να μετακινούνται επειδή έτσι αποφασίζουν οι ίδιοι όπως έκανα εγώ. Όχι από πείνα ή από ανασφάλεια ή από τον κίνδυνο που υφίστανται. Ας απομακρυνθούμε λιγάκι από αυτό το σκεπτικό ότι αν δώσουμε βοήθεια στις αφρικανικές χώρες που είναι η πηγή της μετανάστευσης θα σταματήσουμε αυτήν τη ροή. Ίσως να οδηγούσε σε μια διαφοροποίηση ή σε μια κάποια αντιστάθμιση αλλά συνολικά θα αποτύχει αυτό το τέχνασμα. Τώρα αναφερθήκατε σε κάποιους τομείς, ε, γεωργία, αλία, θα προσέθετα και τη μετανάστευση, είναι βασικό πρόβλημα και νομίζω ότι η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσε και πρέπει να είναι σημαντική εδώ. Παράδειγμα, προσχεδιάζουμε παρεμβάσεις και δράσεις σε διάφορες αφρικανικές χώρες για να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης σε επίπεδο κοινότητας για να μην χρειάζεται οι άνθρωποι να φύγουν. Ταυτόχρονα επιστρέφουμε στις ίδιες αυτές χώρες αδιακρίτως αριθμό μεταναστών χωρίς να υπολογίζουμε κατά πόσο αυτές οι επιστροφές θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο επί των όσων προσπαθούμε να κάνουμε στα πλαίσια της εταιρική σχέσης. Όσο έχουμε τέτοιες αντιφάσεις στην πολιτική μας και στην προσέγγιση μας, μέτρων που θέλουμε να λάβουμε στην εσωτερική διάσταση αφενός και μέτρων που λαμβάνουμε στην εξωτερική διάσταση αφετέρου, θα έχουμε σημαντικότατες αρνητικές συνέπειες όχι μόνο για τις ροές της μετανάστευσης, όχι μόνο για τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων, αλλά για το μέλλον των χωρών μας. Χρειάζεται να λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις διαστάσεις, και την ιστορική και την ιστορική και την ανάπτυξη. Και βεβαίως, όπως έλεγα πριν, υπάρχει δέσμευση των κρατών μελών να μην εφαρμόζει αιρεσιμότητα για να δώσει αναπτυξιακή βοήθεια. Ωστόσο, πολλές από τις ε, μεταναστευτικές μας αποφάσεις ακριβώς τούτο κάνουν. Δίνουν κίνητρα υπό την προϋπόθεση της αποτελεσματικής συνεργασίας στον έλεγχο των ροών. Εδώ χρειαζόμαστε οπωσδήποτε συνέπεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Νκόντο Ντάγκ. Με συγχωρείτε για το πώς ε, πρόφερα το όνομα σας. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε γιατί εσείς μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω ως Πρόεδρος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου με γνώση ε, όλης Αφρικανικής Υπήρου. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να ευχαριστήσω τον πολύ καλό μου φίλο τον Ντανέλ μακάρι με τον οποίο καταφέραμε να επιλύσουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει να κάνει με την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων στην Κεντρική Αφρική. Ξέρετε ότι σε μια συνδιάσκεψη που έγινε πριν από λίγο καιρό αποφασίσαμε να άρουμε τις, τα δασμολογικά εμπόδια τα οποία υφίστανται στην περιοχή εκείνη και που εμπόδιζαν όχι μόνο την κινητικότητα των προϊόντων, αλλά επίσης ε, και την ίδια την κινητικότητα των πολιτών. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της μετανάστευσης, η, Αφρικα... Αφρική σήμερα γνωρίζει δύο είδη μετανάστευσης. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, με απόλυτη ειλικρίνεια. Κυρίως εμείς, οι βουλευτές, έχουμε την εσωτερική μετανάστευση, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι οφείλεται σε κλιματικούς λόγους. Ξέρετε ότι η Αφρική υποφέρει αυτή τη στιγμή από τις κλιματικές αλλαγές. Το Τσάντ, για παράδειγμα, είχαμε δυόμιση, η λίμνη Τσάντ μάλλον, είχε μια τεράστια έκταση στο παρελθόν, αυτή τη στιγμή έχει συρρυκνωθεί. Καταλαβαίνετε ότι όσοι ζούσαν γύρω από τη λίμνη Τσάντ, χρειάστηκε να μεταναστεύσουν. Και βέβαια δημιουργήθηκε ένα κλίμα ανασφάλειας με το φαινόμενο Μπόκο Χαράμα. Καλούμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μεμονωμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσουν. Έχουμε μία κοινή ιστορία. Ξέρετε ότι υπάρχει μια ιστορία που μας συνδέει και θα πρέπει από κοινού να καταφέρουμε να βρούμε προβλήματα τα οποία ταλανίζουν αυτή τη στιγμή την Αφρική. Γι' αυτό το λόγο Σα ζητούμε αυτή τη στιγμή ω ευρωβουλευτέ να ασκήσετε πίεση προκειμένου να εφαρμοστεί η Συμφωνία των Παρισίων και να καταφέρουν να αποφεληθούν οι πολίτε τη Αφρική. Ξέρουμε ότι εξαιτία των κλιματικών αλλαγών έχουμε μια πολύ σημαντική εσωτερική μετανάστευση στην Αφρική, όπω σα το είπα. Πλήττεται επίση η γεωργία μα. Δεν μπορούμε πλέον να ελέγξουμε την αλληλουχία των εποχών, οι οποίες δεν είναι τόσο ξεκάθαρες ω το παρελθόν. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να επωφεληθούμε απλώς από τις ενισχύσεις που μπορείτε να μας δώσετε από κάποιες ευνοϊκές συμφωνίες για γεωργικά προϊόντα τα οποία συνάπτουμε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Εμείς θεωρούσαμε ότι μετά από 20 και πάνω χρόνια διαπραγματεύσεων θα μπορούσαμε επιτέλους να υποφεληθούμε από την ε, Συμφωνία των Παρισίων και ξέρετε ότι στη συνεχεία με τη συνθήκη του Μαρακέ θέλαμε να δώσουμε συνέχεια στι διαπραγματεύσει αυτέ. Δεν μπορούμε να περιμένουμε όμω πλέον να εφαρμοστούν τα συμπεράσματα τη συμφωνία αυτή όταν πλήττονται τόσοι πολλοί πολίτε μα. Στη Λιβύη μπορεί να μην έχουμε πλέον δουλεία επίσημα, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι πολλούνται αυτή τη στιγμή σε τιμή χαμηλότερη από το ζωικό κεφάλαιο οι ίδιοι πολίτε, οι μετανάστε στη χώρα αυτή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γνωρίζουμε πώς ξεκίνησε η κατάσταση στη Λιβύη και ζητάμε από τους Αφρικανούς αυτή τη στιγμή να αναλάβουν δράση. Ποιος ελέγχει αυτό το μη κράτος που είναι η Λιβύη σήμερα. Ξέρετε ότι στο παρελθόν ορισμένοι ήταν τα πράγματα πολύ απλοϊκά λέγοντας ότι έχουμε ένα δικτάτορα και πρέπει να τον βγάλουμε από τη μέση. Ωραία, έγινε αυτό. Τώρα όμω τι κάνουμε. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να βαρύνουν οι ευθύνες μόνο την αφρικανική πλευρά. Από κοινού Αφρικανοί και Ευρωπαίοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αναλάβουν δράση προκειμένου να επιληθεί το πρόβλημα της Λιβύης. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα του εκδημοκρατισμού και λέω εκδημοκρατισμό της Υπήρου γιατί αυτό έγινε, ξέρετε, με έναν τρόπο πολύ γρήγορο με μια συγκεκριμένη αιρεσιμότητα, χωρί όμω να καταφέρουμε τελικά εμεί να προωθήσουμε πολιτικό πλουραλισμό σε όλε τι χώρε. Δύο εθνότητε αυτή τη στιγμή μάχονται στην γένεια. Μπορούμε αυτό να το ονομάσουμε δημοκρατία. Δεν έχουμε καταφέρει εμείς, δεν καταφέραμε να διαμορφώσουμε συγκεκριμένες νοοτροπίες στους εκλογείς μας, δεν καταφέραμε να τους εκπαιδεύσουμε και να τους καταρτήσουμε και μία νυχτή μας λέτε επιβάλλετε εσείς τη δημοκρατία στις χώρες σας. Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό τόσο γρήγορα. Ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν εκατοντάδες πολιτικά κόμματα στην Αφρικανική Ήπειρο χωρίς να έχουν συγκεκριμένη συνειδητή πολιτική ιδεολογία. Και πολύ συχνά, ιδίω από τις χώρες, τις χώρες εκείνες που βγαίνουν από μια σύγκρουση, από μια διένεξη, βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικότητα προβλήματα. Η κατάσταση στη Ζιμπάμπουε τώρα. Ξέρετε ότι αυτοί οι οποίοι έδωσαν αγώνα για την απελευθέρωση είναι τώρα αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να αλλάξουν το καθεστώς. Έχουμε τον ε, επικεφαλής της χώρας, ο οποίος δεν θέλει να εγκαταλείψει την εξουσία, μόλον ότι το ζητούν αυτό πλέον διακαώς οι πολίτες της χώρας. Τώρα, όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το οποίο περιμένουμε από εσά που είστε συνάδελφοί μας, είναι να ασκήσετε πίεση, μεγαλύτερη πίεση ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της μεταφοράς τεχνολογίας. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι υπάρχουν χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκμεταλλεύονται τις πρώτες σύλλες της Υπήρου μου και από την άλλη δεν γίνεται τίποτα προκειμένου να καταφέρουμε να τονώσουμε λίγο περισσότερο την απασχόληση στην Αφρική. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί Αφρικανοί μετανάστες στην Ιταλία για παράδειγμα, οι οποίοι ε, όταν τους ρωτάει κανείς αν θέλετε να επιστρέψετε στην Αφρική λένε μα προφανώ και ναι. Θα πρέπει όμω να μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση στην Αφρική μέσω επενδύσεων. Ξέρετε ότι η μεταναστευτική διαδρομή που ακολουθείται τώρα από του περισσότερου μετανάστε είναι η διαδρομή, ο δρόμο του θανάτου. Το αποκαλέσω, το αποκαλέσω πραγματικά έτσι. Είναι πολλέ φορέ ένα δρόμο χωρί επιστροφή. Αν καταφέρναμε πραγματικά να είχαμε θέσει απασχόληση για του νέου μα, οι οποίοι μπαίνουν όλο και περισσότερο στην αγορά εργασία, θα είχαμε καταφέρει να λύσουμε το ζήτημα τη μετανάστευση. Το σχέδιο Μάρσαλ δεν μπορεί να λειτουργήσει για μια υπορία σαν την, Αφρική, σαν την Αφρική. Χρειαζόμαστε οικονομικό μετασχηματισμό στην Αφρική, εκβιομηχάνηση της Υπήρου και καλύτερη εκμετάλλευση των πρώτων υλών με δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην ίδια την Αφρική όμως. Ο ρόλος τώρα των γυναικών. Εμείς στα πλαίσια του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου έχουμε προωθήσει ως πρώτη μας προτεραιότητα τη θέση των γυναικών. Κάνουμε κάθε το δυνατό προκειμένου να προωθήσουμε περισσότερο τις γυναίκες. Πώς μπορούμε όμως να επιλύσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τις γυναίκες και για τα κορίτσια, αν δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τίποτα στις νέες αυτές γυναίκες οι οποίες θα βγουν στην αγορά εργασίας, αν δεν καταφέρουμε να δώσουμε ένα όραμα για τους νέους μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να καταγγείλουμε καταρχάς αυτά τα οποία γίνονται σήμερα στη Λιβύη, όπου πουλάμε πραγματικά ανθρώπους. Πολύ καλύτερη μοίρα αξίζουν οι κάτοικοι της χώρας αυτής. Και η δεύτερη έκκληση που σας κάνω είναι να καταβάλλετε προσπάθειες προκειμένου η Συμφωνία των Παρισίων να εφαρμοστεί στην πράξη. Ξέρετε ότι ε, θα μπορούσατε εσείς να αναλάβετε συγκεκριμένη δράση ως δυτικές χώρες προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στην Αφρική και ιδίω όσον αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Εμείς σαφώς θα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι, εμείς είμαστε στη διάθεσή σας για να μοιραστούμε μαζί σας τις ευθύνες που μας βαρύνουν, αλλά αντίστοιχη στάση θα πρέπει να υιοθετήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Α μην εθελοτυφλούμε, πρέπει χάρη στην Ευρώπη να καταφέρει και η Αφρική να έχει μια ευκαιρία οικονομική ανάπτυξη. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Μαγκ Μαγκαγκέγκη είναι ο τελευταίο μα ομιλητή. Like to... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Παντσέρη για την δημοκρατία στην Αφρική και την προστασία των ελευθεριών και μίλησε για το πρίσμα των εξελίξεων σε σχέση με την μετανάστευση. Θα ήθελα να αναφερθώ στην παράνομη και όχι την νόμιμη μετανάστευση. Ο συνάδελφος εδώ όταν μίλησε νομίζω είπε ότι η ανάπτυξη δεν είναι πανάκια για το θέμα της ε, μετανάστευσης. Και... Βεβαίως ε, το θέμα είναι ακριβώ ε, και η παράνομη μετανάστευση και ο κύριος Παντσέρη αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Ζιμπάμπουε την ε, Κένια και σε κάποιες αφρικανικές χώρες όπου η δημοκρατία κινδυνεύει. Αλλά οι δύο-τρεις αυτές χώρες ε, ε, δεν προσωπεύουν την Αφρική σήμερα. Μπορούμε οπωσδήποτε να τα πάμε καλύτερα, δεν τίθεται ζήτημα. αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό η δημοκρατία να είναι εθερεωμένη στην Αφρική για να δημιουργηθεί ένα, επιβα... ένα περιβάλλον για άμεσες ξένες επενδύσεις ε, το οποίο επιζητούμε για να υπάρξει ανάπτυξη η οποία θα αποθαρρύνει την παράνομη μετανάστευση για τους επενδυτές όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά για να επενδύσουν οι επενδυτές τα λεφτά τους, σαφώς θέλουν ένα δημοκρατικό πλαίσιο, θέλουν να υπάρχουν νόμοι που θα τηρούνται, εδώ είναι ο δικός μας ο ρόλος ως νομοθέτες, θέλουν μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη που θα επιλύει τις διαφορές και θα προστατεύει οπωσδήποτε τις επενδύσεις τους. Όταν αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανησυχίες, ε, ε, νομίζω θα έχουμε κάνει μεγάλα βήματα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Και Οπωσδήποτε θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα πούμε ε, όλη τη βδομάδα. Είδαμε το... Έχουμε και τη διάσκεψη ψηλού επίπεδου και βεβαίως ε, θα τα πούμε και εκεί. Εγώ δράτω με τις ευκαιρίες ως προεδρεύων αυτής της Επιτροπής να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές μας, τους ε, καλεσμένους μας, τους βουλευτές μας και βεβαίως αναμένω την συνέχεια της εβδομάδας για να είμαστε σε επαφή. Λοιπόν, λίγη η σημερινή μας συνεδρίαση και θα επαναλάβουμε τη συνεδρίαση αύριο στις 9 με την ψηφοφορία. Παρακαλώ λοιπόν να είστε ακριβώς εδώ στις 9. Τα λέμε αύριο. Τελειώσαμε. Καλό σας βράδυ. Καλό ταξίδι.